Okay. Um, good morning everybody and uh, welcome to... Uh, Καλημέρα. Ξεκινάμε αυτή την ακρόαση για την οικονομική κρίση και τη σχέση της με την ε, ισότητα των φίλων. Χαίρο που βλέπω τόσους πολλούς ε, εδώ. Να δώσω το λόγο κατευθείαν στο πρώτο μιλτή ο κύριος Πιτέλα, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και μια σειρά αγοριτών. Παρακαλώ κύριε αντιπρόεδρε. Αγαπητά μέλη, αγαπητέ πρόεδρε, Μάικλ Γκούσταυσον, Μικέλε στα Ιταλικά. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω εξ ονόματος του πρόεδρου κ. Μαρτίν Σούλτς σήμερα σε αυτή την εκδήλωση για την Διεθνή ημέρα των γυναικών. Καλώς ήλθατε, το απευθύνω σε όλους και ιδίως όλες τις γυναίκες στην αίθουσα. Με τιμά που με καλέσετε να ανοίξω την εκδήλωση αυτή σήμερα για την Διεθνή ημέρα των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργανώνει η Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των Φύλων με την υποστήριξη της Διεύθυνσης ε, Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Χαίρο που βλέπω τόσους πολλούς εκπροσώπους Εθνικών Κοινοβουλίων στην ε, αίθουσα αυτή. Μετά την ενίσχυση της ε, θέσης των Εθνικών Κοινοβουλίων μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας, η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια εντάθηκε σημαντικά. Το 2013 η Διεθνής ημέρα γυναικών θα ασχοληθεί με το θέμα η απάντηση των γυναικών στην κρίση. Η εκδήλωση λοιπόν σήμερα θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να συζητήσουν την κατάσταση των γυναικών και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές τέτοιες συζητήσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ισότητας των φύλων που, πρέπει, που τίθενται στο περιθώριο κατά την παρούσα οικονομική κρίση είναι κάτι το αναγκαίο. Όπως γνωρίζετε, το, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει από το 2008 και μετά την ε, βαθύτερη οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση στην ιστορία της από τη δεκαετία 30 και τη Μεγάλη Ήφεση. Αυτό έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους πολίτες της Ένωσης, ιδίως δε στις γυναίκες και την προστασία των δικαιωμάτων τους. Η αύξηση των ποσοστών αντεργίας, η λιτότητα, οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες επηρεάζουν κατά βάση και απευθείας τις γυναίκες επιπλέον. Η κρίση έχει επιδεινώσει τις, ε, τα συμβάντα βίας κατά των γυναικών, την παρενόχληση, τη βία στο χώρο εργασίας ε, και στο σπίτι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση των γυναικών κατά τη διάρκεια της κρίσης και της οικονομικής ύφεσης. Επανέλαβε σε πολλά πρόσφατα ψηφίσματα του ότι είναι ζωτική σημασία να ενισχυθεί η έμφυλη διάσταση και να αντιμετωπιστούν και να βρεθούν μέσα για την αντιμετώπιση και έξοδο της κρίσης. Στις 19 Φεβρουαρίου η Επιτροπή υιοθέτησε ένα, ψήφις, ένα σχέδιο ψηφίσματος σχετικά όπου υπογραμμίζει ότι η οικονομική κρίση έχει διαφοροποιημένο αντίκτυπο στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο στη δεύτερη φάση της κρίσης που χαρακτηρίζεται από περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Συντονισμένη δράση σε επίπεδο ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών με συγκεκριμένα στοχοθετημένα μέτρα για τις γυναίκες απαιτούνται για να αλλάξει η κατάσταση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η κρίση παρέχει την ευκαιρία για να ξανασκεφτούμε και πολιτικές και προτεραιότητες, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε την κρίση ως ευκαιρία για να επιταχύνουμε τις διαθροντικές και κοινωνιακές αλλαγές. Προσβλέπω σε μια καρποφόρα και ζωντανή συζήτηση και σας ευχαριστώ όλους και όλες για το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά σας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πιτέλα. Χαιρόμαστε που είστε σήμερα μαζί μας ε, και μπορείτε να συμμετάσχετε στη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. We'll Ας προχωρήσουμε. για, θεσπίστηκε η η διεθνή ημέρα των γυναικών το Μάρτιο του 1911 στην Αυστρία και πάνω από ένα εκατομμύριο μετήχαν σε εκδηλώσεις για να προωθήσουν την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία η σημερινή ημέρα για να γίνει ένας πολιτικός διάλογος στο Κοινοβούλιο για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις γυναίκες. Επίσης μπορούμε έτσι να κοινοποιήσουμε ε, τα όσα κάνει το Κοινοβούλιο στους πολίτες ε, και δεδομένης ε, της τωρινής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη Έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε παρουσία του Αντιπροέδρου Πιτέλα, ε, τις επιπτώσεις που έχει αυτή η σοβαρότατη κρίση ε, για την κατάσταση των γυναικών και να διερευνήσουμε ε, πιθανές λύσεις για την έξοδο από την κρίση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους, τα μέλη του πρώτου αλλά και του δεύτερου πάνελ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεχτήκατε τη σημερινή μας πρόσκληση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μογάν Σαρτιέ για την παρουσία της. Είναι η συγγήτρια για μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση ε, που εγκρίθηκε τους περασμένους μήνες στην Επιτροπή Γυναικών και που θα ψηφιστεί και στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Μας προσέφερε μια ολιστική προσέγγιση για το σύνολο των επιπτώσεων της οικονομικής ε, ύφεσης επί των γυναικών και εξέφρασε πολύ ενδιαφέρουσες ε, θέσεις σε σχέση με ε, πιθανές ε, λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη το ζητούμενο, δηλαδή την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ο κύριος Άντελ δεν μπορεί δυστυχώς να έρθει σήμερα, αλλά θα αντικατασταθεί από πρόσωπε Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, ο Επίτροπος θα έχει ηχογραφήσει, μαγνητοσκοπήσει ένα μήνυμα, το οποίο θα παρακολουθήσουμε στην συνέχεια. χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι αθρώη προσέλευση των ομολόγων μας από τα κράτη-μέλη. Ε, με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ένα αυξημένο ρόλο στην ε, ευρωπαϊκή νομοτεχνική διαδικασία για την αναθεώρηση των πρωτοκόλων 1 και 2 της συνθήκης. Ο πολιτικός διάλογος ενισχύθηκε ε, ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν το, την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας μέσα από ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση, ένας τακτικός διάλογος ανάμεσα ε, στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι υψίστης της ε, σημασίας ε, και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που θα σημάνω τώρα την έναρξη του πρώτου διαλόγου για τις επιπτώσεις κρίσης επί των γυναικών και τις μελλοντικές προοπτικές για τις γυναίκες. Προτού περάσουμε στο πρώτο πάνελ θα ήθελα να σας πω κάποιες πρακτικές πληροφορίες και θα περάσω στα Σουηδικά γιατί είναι πιο εύκολο για μένα. Εάν ε, αν δεν καταλαβαίνετε Σουηδικά θα σας πρότεινα να βάλετε ακουστικά γιατί αλλιώς δεν θα με καταλάβετε. Den, den här dagen um, Έχουμε την οργανώσει τη συζήτησή μας σε τρία τμήματα. Και μετά από κάθε πάνελ θα έχουμε έρωτα απαντήσεις ε, για να υπάρξει ανταλλαγή με τα μέλη του πάνελ. Το πρώτο τμήμα είναι πολύ συντομότερο σε σχέση με τα άλλα δύο. Ε, δεν θέλουμε να κάνουμε μακροσκελέστατες ε, παρεμβάσεις. Ε, μας ενδιαφέρουν οι ερωτήσεις που θα απευθύνεται στα μέλη του πάνελ. Θα είναι κατά τι μακρύτερο το δεύτερο τμήμα. Ε, έκαστος μπορεί να έχει τρία λεπτά στη διάθεσή του για να παρέμβει και μπορείτε να κάνετε και επερωτήσεις. Μπορούμε να κάνουμε τέσσερις, πέντε ερωτήσεις ε, τη φορά και στη συνέχεια να οργανώνουμε δεύτερο, τρίτο γύρο ερωταπαντήσεων. Για να ε, μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το σύστημα όπως το έχουμε προβλέψει θα πρέπει να συμπληρώσετε το δελτίο για το αγόρευσης που σας έχουμε διανύμει για να εγγραφείτε στον κατάλογο ομιλητών και να σας δώσουμε το λόγο στη συνέχεια. Νομίζω ότι δεν έχω κάποιες άλλες ε, πρακτικού χαρακτήρα πληροφορίες για να σας δώσω και μπορούμε να αρχίσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ε, βλέπω σήμερα. Θα, αρχίσουμε με τη σειρά. Πρώτη θα πάρει το λόγο η κυρία Σίλβια Βουάλμπι, που είναι καθηγήτρια Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Έχετε στη διάθεσή σα 10 λεπτά για την αγορευσή σου. Παρακαλώ. I'm here Καλημέρα Σήμερα βρίσκομαι μαζί σας για να μιλήσω για την δημοσιονομική και οικονομική κρίση και την αντίδραση των γυναικών σε αυτήν. Θα μιλήσω γι' αυτό αναφερόμενοι σε πέντε σημαντικά σημεία. Θα συζητήσουμε τη σχέση των ε, εμφυλοποιημένων αποφάσεων, της ανισότητας του αντικτύπου της κρίσης σε άντρες και γυναίκες, τους εμφυλοποιημένους ε, τρόπους αντιμετώπισης των δημοσιονομικών ελλημάτων στις ε, στρατηγικές και τέλος στην συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, το mainstreaming. Καταρχάς, η λήψη αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα είναι κυρίως από άνδρες. Ασχολείται, μάλλον, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της κοινωνικής ζωής, ο οποίος επηρεάζει όλους. εκείνοι που επηρεάζονται από τον τομέα αυτό πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες πρέπει να εκπροσωπούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα, διότι δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα, είναι δημόσιο το ζήτημα και αφορά όλους. θεωρούμε πως η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι βελτιωμένη όταν συμπεριλαμβάνονται και οι γυναίκες. Μειώνεται ο, το ρίσκο στην ε, λήψη αποφάσεων. Η ύφεση τώρα. Πολλαπλές υφέσεις παρατηρείται μία... Ε, παρατηρείται άνισος αντίκτυπος της κρίσης σε άντρες και γυναίκες. Στην αρχή οι άντρε ήταν εκείνοι που επηρεάστηκαν δυσανάλογα διότι η κρίση επηρέασε τον κατασκευαστικό τομέα. Υπήρχε διαχωρισμό βιομηχανικό, δηλαδή η διαφορετική κλάδοι τη βιομηχανία επηρεάστηκαν διαφορετικά και επίσης και άντρε και γυναίκες που εργάζονται σε αυτή. Έπειτα, η κρίση επηρέασε δυσανάλογα τις γυναίκες διότι οι περικοπές στα δημόσιες δαπάνες επηρέασαν με τη σειρά τους δυσανάλογα τομείς της οικονομίας στους οποίους απασχολούνται κυρίως γυναίκες. Στον τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα, στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της περίθαλψης και των υπηρεσιών αποτροπής της βίας ενάντια στις γυναίκες. Και εκεί έγιναν περικοπές, καθώς και σε άλλες δημόσιες δαπάνες. Έτσι λοιπόν η έμφυλη διάσταση της κρίσης είναι άνηση και επηρεάζεται από τη φύση της ε, αντίδρασης των κυβερνήσεων στην κρίση. Υπάρχουν επιλογές ως προς την πολιτική και την, ε, για την αντιμετώπιση της κρίσης, διαφορετικές σε άντρες και σε γυναίκες. Πολλές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πίεση για τη μείωση του δημοσιονομικού του ελλείμματος. Δεν θα σας ε, μιλήσω για, και θα επιχειρηματολογήσω για το αν θα πρέπει να ε, μειωθεί αυτό και το πώς πρέπει να γίνει, αλλά για το πώς μειώνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτή η επιλογή είναι έντονα αμφιλοποιημένη. Τα ελλείμματα μπορούν να περικοπούν είτε αυξάνοντας τους φόρους, είτε περικόπτοντας τις δημόσιες δαπάνες. Όταν αυξάνονται οι φόροι, εκείνοι αφορούν κυρίως τους άντρες, είτε με την ε, διαφορετική αντιμετώπιση των φορολογικών ε, παραδείσων, είτε με την καταπολέμηση της φοροαποφυγής πολλές χώρες αποφάσισαν να περικόψουν τις δημόσιες δαπάνες από την άλλη. Και η επιλογή αυτή, έναντι, ε, αντί για την αύξηση των φόρων, είναι μια εμφυλοποιημένη επιλογή και οδήγησε σε δυσανάλογα άσχημο αντίκτυπο εις βάρος των γυναικών. Ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών, όπου χρησιμοποιείται κυρίως από γυναίκες. Στους τομείς που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης, η φορολογία είναι εμφυλοποιημένο ζήτημα. Η κατάρτιση εμφυλοποιημένου προϋπολογισμού είναι μια τεχνική η οποία μας δείχνει το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι εναλλακτικές στρατηγικές ε, μείωσης του ελλείμματος είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της συνεκτίμησης της διάστασης ε, του φύλου στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, ε, τρόποι εξόδου από την κρίση. Ας μην κοιτάζουμε πίσω σε αυτά που έγιναν και σε αυτά που γίνονται, αλλά ας κοιτάξουμε επίσης και προς το μέλλον. Η στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης έχει και αυτή εμφυλή διάσταση. Έχουμε πολλές επιλογές ως προς τον τρόπο που θα επιτύχουμε την οικονομική ανάπτυξη. Και οι επιλογές αυτές έχουν επίσης έμφυλη διάσταση. Ίσως περισσότερο από άλλους τομείς. Η ενίσχυση της ε, συμμετοχής των γυναικών έχει πολύ μεγάλη σημασία στην μείωση της ε, ανεργίας μέσω πολιτικών που μπορούν να συμφιλιώσουν την ε, οικογένεια και την εργασία, μέσω πολιτικών που ενθαρρύνουν την πλήρη απασχόληση των γυναικών και την μέγιστη παραγωγικότητά τους προς όφελος της οικονομίας. Αυτή ήταν η παραδοσιακή οδός που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχει την οικονομική ανάπτυξη. Έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν εναλλακτικέ στρατηγικές για την οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα η στρατηγική της απορρίθμισης. η απορρίθμιση ερμηνεύεται πολλές φορές ε, μόνο ως η απομάκρυνση της ε, υπερβολικής γραφειοκρατίας. Αλλά πολλές φορές αυτό οδηγεί σε μείωση τη ανεργία και αύξηση της απασχόλησης με την ε, ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Επίσης, παρέχονται οι δυνατότητε στις γυναίκες να ε, έχουν απασχόληση, δίνοντας στις γυναίκες πρόσβαση σε άδειες μητρότητα, σε επιδόματα μητρότητα και σε θέσεις απασχόλησης στον τομέα της ε, περίφευξης και της φροντίδας. Οι γυναίκες συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη και είναι μέρος της θετικής οικονομικής ανάπτυξης. Έχουμε προτείνει για να βγούμε από την ε, κρίση να γίνουν επενδύσεις. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ε, όπου μπορούν να γίνουν επενδύσεις και αυτοί έχουν έμφυλη διάσταση. Εάν επενδύσουμε σε μια οικονομία γνώσεων, όπως έχει προτείνει στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα περιλαμβάνει την συμπερίληψη των γυναικών στην οικονομική στρατηγική για την αύξηση της παραγωγικότητας. Πολλές φορές όμως παρατηρήθηκε ε, για την αντιμετώπιση της κρίσης μια μεταστροφή στις παραδοσιακές μορφές βιομηχανίας. Για παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών παρατηρήθηκε επιστροφή στις παραδοσιακές μεθόδους μεταφοράς και αυτό έχει έμφυλη διάσταση, διότι οι άνδρες υπερεκπροσωπούνται στον τομέα των μεταφορών. Παρατηρούμε επομένως έναν έντονο διαχωρισμό εις βάρος των γυναικών στην βιομηχανία και στις μεταφορές. Τώρα, οι στρατηγικές για την ανάπτυξη θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ε, συμπερίληψη, περισσότερη συμπερίληψη των γυναικών και καλύτερες υποδομές ε, για μια στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης. Έχουν γίνει έλεγχοι και μελέτες αντικτύπου, οι οποίε έχουν δείξει την έντονα έμφυλη διάσταση. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε και επιθυμούμε να συνεχίσουμε την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και το εφαρμόσουμε αυτό στην οικονομία, θα δούμε ότι ενώ έχει εφαρμοστεί με επιτυχία για την αντιμετώπιση της φτώχειας, δεν είχε την ίδια επιτυχία εφαρμογή σε ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης. έχουμε επιτύχει μία ίση εκπροσώπηση των φίλων στον τομέα της δικαιοσύνης. Όμως άλλοι τομείς της οικονομίας δεν είχαν τόσο θετικά αποτελέσματα και τόσο καλή εφαρμογή. Η συνεκτίμηση λοιπόν της διάστασης του φίλου μπορεί να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της άνησης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στην οικονομία. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, η δημοσιονομική και η οικονομική κρίση έχει έμφυλη διάσταση, έχει αιτίες και έχει επιπτώσεις. Η έμφυλη διάσταση της ε, χαράξης πολιτικής οδήγησε στα άνισα αποτελέσματα της κρίσης στις επιπτώσεις, ανητικές επιπτώσεις στις γυναίκες, όμως έχουμε την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε την ε, τακτική για την οικονομική ανάπτυξη ως προς ε, τα δύο φύλλα και να την εφαρμόσουμε. Να εφαρμόσουμε τις τεχνικές λοιπόν του mainstreaming στην ε, χάραξη δημοσιονομικής πολιτικής έτσι ώστε να επιτύχουμε ταυτόχρονα και οικονομική ανάπτυξη και ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ευχαριστώ. Eh, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θέλω να μιλήσω σου ειδικά παρακαλώ τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστούμε διότι καταδείξατε με σαφήνεια ότι όταν μιλάμε για στατιστικά στοιχεία, και ε, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές για να εκφράσουμε την πραγματικότητα, πάντοτε υπάρχει χώρος για να εξετάσουμε το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια Σαλομέ Μπουγκούα, Γενική Διευθύντρια του Ακίντουα, Εθνικό Σύνδεσμος Μεταναστριών στην Ιρλανδία. Δέκα λεπτά έχετε κι εσείς στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα σήμερα εδώ και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας των δύο φίλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με προσκάλεσε στην σημερινή συνεδρίαση. Είμαι από την Ιρλανδία όπως ακούσατε και εργάζομαι στο δίκτυο, στο σύνδεσμο μεταναστριών ε, στην Ιρλανδία αλλά είμαι και πρόεδρος ε, των, ε, της Ένωσης Μεταναστριών στην Ιρλανδία που συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Λόμπι εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, θα ήθελα να ε, εκφράσω τις απόψεις των μεταναστριών που εκπροσωπώ. Ας αρχίσω λοιπόν την παρέμβασή μου. Η τωρινή παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση δημιουργεί ε, πάρα πολύ σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις ε, και για τα δύο φύλλα ανά τον κόσμο, αλλά πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες διότι είναι πολύ χαμηλότερη η μισθή τους. 22% είναι η διαφορά στους, η μισθολογική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα και χάνουν πρώτε τη δουλειά τους ε, σε περιόδους ε, κρίσης. Ε, αναμφισβήτητα λοιπόν ήταν αρνητικές οι επιπτώσεις για τις γυναίκες, η υψηλότερη ανεργία, μειωμένη πρόσβαση στους πόρους και πτώχευση των γυναικών σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων διότι οι γυναίκες ολόκληρο τον κόσμο εργάζονται επί πλήστο στη μεταποιητική βιομηχανία ε, και ε, εργάζονται στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, ή κοινωνικής περίθαλψης, περίθαλψη ηλικιωμένων και παιδιών και νομίζω ότι γι' αυτό πλήττονται περισσότερο οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο λοιπόν από την δική μας ε, προοπτική και επειδή εκπροσωπώ τις μετανάστριες ε, έχω ήδη όμως διαπιστώσει ότι η αυξανόμενη ανεργία επηρεάζει τη ιδιαίτερως ε, τις μετανάστριες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν ή δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να έχουν πρόσβαση στους απαιτούμενους πόρους και αυτό επηρεάζει αυξήσει την ικανότητά τους ε, να ε, καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες ε, των παιδιών και της οικογένειάς τους. Από το 2008 στο 2013, κατά τη διάρκεια δηλαδή της Ιρλανδικής χρηματοπιστωτικής κρίσης που απορρέει από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 2007 και 2008, είναι εν μέρη υπεύθυνη για το ότι βούλεξε στην ύφεση η χώρα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ε, ο συνασπισμός Φιάννα Γκέιλ και Πρασίνου Κόμματος ανακοίνωσε επίσημα τότε ότι εισήλθε στην ύφεση η χώρα ε, και αυξήθηκε κατακόρυφα η ανεργία και ήταν η πρώτη χώρα της ζώνης Ευρώ που εισήλθε στην ύφεση βάσει του κεντρικού της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ε, το 2007 και το 2008 ξεκίνησε αυτή η τάση Ε, με δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι 54% το ποσοστό ανεργίας ε, των ε, μεταναστριών γυναικών κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί από το 2001 δηλαδή που απέχουμε από τους στόχους της στρατηγικής 2020 βλέπουμε επίσης το 2002 ήταν 40,7% η ανεργία των γυναικών αυξήθηκε κατά αυξήθηκε ε, κατά κόρυφα το 2009 και τα τελευταία δύο χρόνια, το 2011 έφτασε το 10,1%. Επηρεάστηκε λοιπόν η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά όχι μόνο αυτό. Ε, πλήττονται από ένα φάσμα μέτρων που έχουν αναλυφθεί από μεγάλες επιχειρήσεις. Παραδείγματο χάρη, αποζημίωση για την άδεια μητρότητας. Ένας εκπρόσωπος συνδικαλιστικής οργάνωση είπε ότι υπάρχουν και αυξημένες παρενοχλήσεις των γυναικών στο χώρο εργασίας λόγω της κρίσης. Επίσης, περικοπές ε, των θέσεων απασχόλησης στο δημόσιο τομέα επηρεάζουν ε, περισσότερο τις γυναίκες ε, γιατί εργάζονται στον τομέα υγείας και παιδείας και έτσι οδηγηθήκαμε σε μεγάλη απώλεια θέσεων απασχόλησης και θέσεις διαθεσιμότητα των γυναικών. Λόγω αυτών των δεδομένων, οι γυναίκες θεωρούν ότι δεν είναι ισότιμη πρόσβαση των γυναικών γυναικών στην αγορά εργασίας και στη, ε, ε, κρίνουν λοιπόν ότι λόγω των νέων μέτρων που λαμβάνονται υφίστανται με ε, διακριτική μεταχείριση. Βάσει στατιστικών στοιχείων βλέπουμε ότι ο αριθμός ανεργία, ε, ο, το, το ποσοστό ανεργίας για τους μετανάστες είναι 22% κατά τη διαστολή με το ποσοστό ανεργίας στην Ιρλανδία που είναι 18,5%. Ε, υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και τίθεται ζήτημα ενσωμάτωσης αυτών των γυναικών και των παιδιών τους στην κοινωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ιρλανδία βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της κρίσης. Σε πολλές ε, οικογένειες ζουν με το μισθό της γυναίκας που είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Ε, παλεύουν οι γυναίκες να ε, καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και ένα τέταρτο των οικοκυριών δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν συνάψει ε, επίσης υπάρχει μειωμένη υποστηρίξη προς τις κοινότητες αυτών των γυναικών στην Ιρλανδία. Οι γυναίκες λοιπόν ε, χρειάστηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης να διακόψουν ε, τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Το ίδιο συμβαίνει και στις ενώσεις που υποστηρίζουν τις γυναίκες. Εμείς παραδείγματος χάρη δεν λαμβάνουμε καμία χρηματοδότηση από το κράτος και έχουμε χάσει και τέσσερα μέλη του προσωπικού μας λόγω των ε, περικοπών. Ε, ε, το πρόβλημα γίνεται όξι διότι κάποιες γυναίκες υφίστανται μέχρι και βία και χρειάζονται την διαρκή υποστηρίξή μας στη συνέχεια. Οι επιχειρήσεις θέλουν να εξοικονομούν χρήματα και στοχοποιούν τις γυναίκες κυρίως ως προς την αποζημίωση για την άδεια μητρότητας. το 2010 λάβαμε πάρα πολλές σε καταγγελίες σε σχέση με τη μειωμένη πρόσβαση στην απασχόληση. Αυξάνεται και η φτώχεια των γυναικών 98% των μονογονεϊκών ε, οικογενειών ε, είναι ανήπαντρες γυναίκες ε, με τα παιδιά τους. Οι μετανάστριες γυναίκες είχαν αρχικά μια άδεια εργασίας και συνέχεια απέκτησαν άδεια διαμονής, αλλά χρειάστηκε να απομακρύνθηκαν μάλλον από την αγορά εργασίας λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, λόγω της κρίσης. Κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις οι μετανάστριες παίρνουν ε, ε, πολύ χαμηλούς μισθούς ε, και οι ανατολικοευρωπαίες μετανάστριες είναι τα σοβαρότερα θύματα αυτής της κρίσης. Άρα βρίσκονται σε επισφαλή θέση και τα υπηρεσίες εξέβρεση εργασίας προσφέρουν ιδιαίτερα επισφαλή θέσεις εργασίας αυτής της γυναίκες. Υπάρχουν περικοπές στις κρατικές παροχές όπως παραδείγματο χάρη μαθήματα γλυκών, αποζημίωση για την περίθαλψη των παιδιών και ούτω καθεξής. Αυξημένος ανταγωνισμός μας οδήγησε επίσης σε περισσότερα επεισόδια ρατσισμού που επηρεάζουν και πάλι περισσότερο τις μετανάστριες. Είναι μεγάλη πρόκληση η ανατροφή των παιδιών για τις μετανάστριες διότι δεν έχουν ρευστότητα και καμιά υποστήριξη από, από την ευρύτερη οικογένεια. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες προτάσεις σήμερα, τέσσερις συγκεκριμένα. Μια ξεκάθαρη έμφυλη στρατηγική με προγράμματα υποστήριξης απασχόλησης χρειάζεται για να κρατήσουν αυτές οι γυναίκες τη δουλειά τους με τη σωστή υποστήριξη, κατάρτιση, επιμόρφωση και την κατάλληλη εμπειρία στην αγορά εργασίας ούτω ώστε να διαδραματίσουν ένα ζωτικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ιρλανδίας. Είναι από τις επαθέστερες κοινωνικές ομάδες μετανάστριες. Επίσης, Επίσης χρειαζόμαστε ένα καινοτόμο κράτος πρόνοιας και στρατηγικές ώστε να, ε, γίνει, να καταρτιστούν έμφυλες ε, πολιτικές ε, και να προσαρμοστούν στις ανάγκες αυτών των γυναικών. Επίσης η Εθνική Στρατηγική για τις Γυναίκες 2007 ως 2016 θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. Στη συνέχεια χρειάζεται μια διαδικασία διαβούλευσης με τις γυναίκες και κυρίως με αυτές τις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες με τρόπο ώστε σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και όσου καταρτίζουν τι πολιτικέ να βρεθούν λύσει για να μειωθούν οι βαθύτερε επιπτώσει τη κρίση στι γυναίκε και τα παιδιά του. Eh, ε, σα ευχαριστούμε για την παρεμβάσή σα. Παρότι λέμε ότι επηρεάζονται περισσότερο οι γυναίκες από την κρίση σε σχέση με τις, τους άντρες αληθεύει, όπως σωστά είπατε, ότι υφίστανται και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως παραδείγματο χάρη μετανάστες που πλήττονται ακόμη περισσότερο, δηλαδή εξορισμού είναι ευπαθέστερες αυτές οι οι ομάδες ε, διότι δεν ενσωματώνονται στην κοινωνία κυρίως ε, κατά την περίοδο αυτή ε, όπου βιώνουμε μια βαθύτατη κρίση. Σας ευχαριστούμε για τις προτάσεις σας. Θα συνεχίσουμε τώρα και θα ακούσουμε την κυρία Σάσα Μπεζουχάνοβα από τη Χιούλετ Packard, Διευθύντρια Αρμόδια για το Δημόσιο Τομέα σε Αναπτυσσόμενες Αγορές και πρόεδρο του Βουλγαρικού Κέντρου για τις Γυναίκες στις Τεχνολογίες. 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Με PowerPoint θα δουλέψω. Οπότε θέλω μια τεχνική υποστήριξη. αισθάνομαι πραγματική τιμή που παρουσιάζω τις απόψεις μου για το θέμα της επίτευξης ισότητας των φίλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από μια άλλη οπτική ωστόσο ως ένα άτομο που μεγάλωσε και εργάζεται επαγγελματικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον σε έναν από τους κλάδους που απαιτούν περισσότερη ένταση γνώσης που είναι η τεχνολογία της πληροφορίας. Θα χρησιμοποιήσω το χρόνο μου προσπαθώντας να σας δείξω κάποιες πιθανές λύσεις για το πώς ε, μπορούμε να καλύψουμε την υφιστάμενη δύσκολη κατάσταση. Δεν δουλεύει η παρουσίασή μου. παρούσα κατάσταση δεν εκπλήσει το ότι υπάρχουν, υπάρχουν μάλλον πολλές στατιστικές για το πώς η φυστάμενη κατάσταση και η κρίση ιδίω επηρέασε την οικονομία της Ευρώπης και του κόσμου. Επιτρέψτε μου να το δω από μια μεγαλύτερη οπτική. Η κρίση προκλήθηκε διότι οι παλιές έννοιες δεν αλλάζουν σε πολλές πτυχές. Βλέπουμε μια ανεργία που δεν έχει προηγούμενο σήμερα. Πάνω από 26 εκατομμύρια άτομα, λένε οι τελευταίες στατιστικές, είναι άστεγοι, μετανάστες, αλλά και εργαζό, παγιοί εργαζόμενοι. Βλέπουμε επίσης ότι τα μοντέλα, τα παγκόσμια οικονομικά μοντέλα αποδεικνύονται ανεπαρκή. Διότι ο στόχος είναι να δώσουν κέρδη στους μετόχους, κάτι που οδήγησε σε, σε μεγάλη χρηματοοικονομική μηχανική που οδήγησε σε και στο σύστημα. Πολλές επιχειρήσεις πλήρωσαν το τίμημα διότι δεν ήταν ε, πλέον να παράσχουν καινοτόμες λύσεις ενώ τρώγαν το χρόνο τους προσπαθώντας να ισορροπήσουν ε, στο εσωτερικό τους διάφορες κουλτούρες. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μετακίνηση του, του, του δυναμικού μας σε χώρες νέες. Πολλοί Ευρωπαίοι φεύγουν στην Νότια Αμερική, στην Ασία, ακριβώς γιατί εκεί βρίσκουν καλύτερες ευκαιρίες εργασίας. Η Ευρώπη χάνει την ανταγωνιστικότητά της γιατί δεν εκμεταλλεύεται τα προσόντα των ανθρώπων αυτών. Μια άλλη διάσταση του θέματος είναι ότι υπάρχει ένα νέο παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Άρα εμφανίζονται νέοι παίκτες στη διεθνή σκηνή. Οι χώρες BRIC, Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία και Κίνα. Όλο ένα και παίζουν αυξανόμενο ρόλο στην διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης της παγκόσμιας οικονομίας η λειτουργία, ο συντονιστικό ρόλος των Ευρωπαίων λοιπόν στη δικασία αυτή αλλάζει. Και το γεγονός ότι η Ευρώπη, η οικονομική κρίση στην Ευρώπη στηρίζεται και προσπαθεί να αντιμετωπιστεί μέσα σε ένα εθνοκεντρικό πλαίσιο κατά βάση, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της γνώσης και των προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με μια αντίστοιχη ανταγωνιστική ατζέντα. Προφανώς υπάρχει και ένα νέο κέντρο που επηρεάζει τις οικονομικές διαδικασίες. Η αστάθεια και οι εξεγέσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική για να μην μιλήσουμε για την αστάθεια που προκαλεί στις ευρωπαϊκές χώρες η οικονομική, το οικονομική κρίση. Η Ένωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε, συγγνώμη, που ήταν καλός και στέρεος εταίρος της Ευρώπης στο παρελθόν, έχει εσωτερικά προβλήματα και δεν ασχολείται τόσο με τη βοήθεια της Ευρώπης. Η Ευρώπη σήμερα δεν έχει επαρκή μοντέλα ή πρόκληση για να ανταποκριθεί στην ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται. Έχουμε έναν γυράσκοντα πληθυσμό μέχρι το 2000 ε, μέχρι το 2020 το ποσοστό των άνω των 65 θα αυξηθεί σημαντικά. Ενώ στον κλάδο μας, πούμε, στα, στην ε, τεχνολογία της πληροφορικής έχουμε ελλείψεις ε, σε ανθρώπινο δυναμικό. Τα νέα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι μέχρι το 2015 θα χρειαστούμε 750.000 νέε θέσει εργασία στον τομέα του, της πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα οι δικοί μας φεύγουν. Πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα αυτό, ποιες λύσεις υπάρχουν, Προφανώς χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τις υφιστάμενες μεθόδους μπορούν να επηρεάσουν την ε, γενικότερη ανάπτυξη. Προφανώ μια καλή εκπαίδευση που στηρίζεται και στο διαδίκτυο είναι ο καλύτερο τρόπος. Ε, τα προσόντα αυτά πρέπει να, να, να παρέχονται χωρίς περιορισμούς και να λαμβάνονται από τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Και αυτό είναι ένα έμφυλο θέμα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα παράσχει ασφάλεια, διαφάνεια και ασφάλεια σε επιχειρήσεις αποτελεί δε έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε και την αποδοτικότητα και την ε, τεχνολογική ανάπτυξη. Επίσης, ο τρόπος που κυβερνιέται μια χώρα, η ηλεκτρονική δημοκρατία, όπως την λέω εγώ, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα ούτως ώστε να προωθήσουμε θέματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία των πολιτών, τη δημοκρατία σε, ένα, μια ευρύτερη διαβούλευση και να ενισχύσουμε την εμπλοκή των πολιτών και την πεποίθησή τους ότι μετέχουν στη λήψη των σημαντικών πολιτικών είτε εθνικών είτε ευρωπαϊκών θεμάτων. Ένα άλλο, μια άλλη σημαντική διάσταση είναι να δουλέψουμε με στόχο την ανάπτυξη νέων προσώνων σε όλο τον πληθυσμό, υπογραμμίζοντας την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα. Αν θέλουμε αύριο να έχουμε μια ανταγωνιστική Ευρώπη, θα έπρεπε να επανεξετάσουμε το πώς διαμορφώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, να ενισχύσουμε τις ιδέες και να προετοιμάσουμε τους πολίτες μας για να αναλάβουν μια ευθύνη για τη δική τους ζωή και να χτίσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ούτως ώστε να έχουν ανταγωνιστικότητα και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ένα αποθεματικό που δεν χρησιμοποιούμε και μπορεί να βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διευρωπαϊκές προκλήσεις είναι, είναι να κινητοποιήσουμε περισσότερες γυναίκες. Αν μπορείτε να δείξετε τα στατιστικά τώρα. Η Μακέντζη ακολουθεί τη θεματική για την ισότητα των γυναικών και την εμπλοκή τους εδώ και δέκα χρόνια σχεδόν. Μαζί με τη Eurostat το χωρίσανε σε μία προβολή για την κινητοποίηση των γυναικών σε επαγγελματικέ αυτές δραστηριότητε. Στο γράφημα αυτό βλέπετε ότι αν μέχρι το 2025 οι μισές από τις κοπέλες ε, που τελειώνουν το σχολείο, ε, το πανεπιστήμιο, μπουν στην ενεργή επαγγελματική ζωή στην ε, ευρωπαϊκή κοινωνία, η απόκληση, το κενό που θα ήταν 21 εκατομμύρια, ε, το, η έλλειμμα, το 21 εκατομμυρίων ε, εργαζομένων με γνώση θα μειωθεί στα τρία. Αν δεν κάνουμε κάτι δηλαδή σε 15 χρόνια θα έχουμε 21 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, που δεν θα μπορούμε να καλύψουμε. Αν από τις, μισέ μισές μόνο οι γυναίκες που τελειώνουν σχολείο και πανεπιστήμιο, ήδη το κενό θα είναι 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια είναι κάτι που μπορείς να το αντιμετωπίσεις με πολλά μέτρα, κινητοποιώντας ε, την τεχνολογία, δημιουργώντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην παραγωγή, με δημιουργώντας νέα μοντέλα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν που ξεπερνά την ε, ψυχολογική ανακούφιση των γυναικών σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και σχετίζεται με, την, ε, με το μέλλον του κόσμου. Έχουμε λοιπόν, γιατί έχουμε για να σας μιλήσω εδώ, γιατί κυρίως θέλω να δω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας να είμαστε επιτυχείς και να μοιραζόμαστε κοινές επιτυχίες, όχι κοινά προβλήματα. Κάποιες από τις καλές πρακτικές προέρχονται από τις ε, παγκόσμιες εταιρείες. Θα σας πω κάποιες από κάποια παραδείγματα για το πώς η κυβέρνηση μου, η Hewlett Packard, ενθαρρύνει την εμπλοκή των γυναικών στην απασχόληση. Η Hewlett Packard απασχολεί 30,7% των γυναικών 30% των υπαλλήλων της είναι γυναίκες. Ένα καλό νούμερο για το χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορίας. Μου λένε οι οργανωτές ε, ότι πρέπει να τελειώσω. Αυτό που κάνουμε είναι να επιτρέπουμε να δουλεύουν ε, από το σπίτι όλοι, όχι μόνο οι γυναίκες. Το 80% των ε, εργαζομένων σε εμά μπορεί να επιλέξουν να δουλεύουν από το σπίτι τους. Οπότε μπορεί μαζί να δουλέψουν από το σπίτι, να ασχοληθούν με την οικογένειά τους και αυτός είναι ο τρόπος να αυξηθεί η επαγγελματική καριέρα των γυναικών. Έχουμε γυναίκες που δουλεύουν σε, που ανταλλάσσουν ε, ε, πληροφορίες και βέλτιες πρακιστίες σε παγκόσμιο επίπεδο για να καταλάβουν τα νέα ζητήματα. Έχουμε προγράμματα ε, μέντορος, ακόμα και σε επίπεδα εκτελεστικού για να βοηθήσουμε γυναίκες. Μια πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για το Βουλγαρικό συγγνώμη, Κέντρο για τις γυναίκες στη τεχνολογία. Αυτό που κάναμε για τη Βουλγαρία και βλέπετε στο γράφημα είναι να εξασφαλίσουμε προγράμματα μοντελοποίησης ρόλων και παροχής μεντόρων σε κάθε επίπεδο από το σχολείο όπου τα κορίτσια εκπαιδεύουν, διαμορφώνουν την άποψή τους για την επιλογή της δουλειάς τους και όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, περιορισμοί ή προκαταλήψεις, ότι ας πούμε μηχανικοί ή πληροφορικάροι είναι άντρες και ε, αυτά τα στερεότυπα προέρχονται από την οικογένεια, από την κοινωνία, αντιμετωπίζονται εισάγουμε βέλτιες πρακτικές, ξεκινούμε αλλαγή νοοτροπίας, υποβάλλουμε στα παιδιά, στα κορίτσια, στις φοιτήτριες, στους νέους επαγγελματίες, ε, ανθρώπους που δουλεύουν στην καριέρα, που θέλουν να διαλέξουν και αν θέλετε μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες σε άλλο επίπεδο. Αυτό το, αυτό το μοντέλο, το, την έννοια του μοντέλου και την έννοια του μέντορα την παρέχουμε σε κάθε επίπεδο. Επίσης δεν δουλεύουμε μόνο με κοπέλες, δουλεύουμε και με αγόρια, γιατί και τα αγόρια πρέπει να αλλάξουν θετικά την οτροπία τους. Παρέχουμε online training ε, και για επιχειρηματίες και για εκπαίδευση στο δίκτυό μα. Το δίκτυο περιλαμβάνει γυναίκες, λίγους άντρε, ανοιχτό είναι πάντως, καλούνται οι άντρε. από τέσσερις διαφορετικές γενναίες ενώ έχουμε και σε επίπεδο sponsoring άνδρες που είναι ηγέτες στην διαχείριση των επιχειρήσεων της χώρας αλλά και παρέχουν τις βέλτιστες σχετικές έννοιες στην επιχειρηματική κοινότητα. Κλείνοντας, εγώ θεωρώ ότι η κρίση της Ευρώπης θα ξεπεραστεί. Αλλά αυτό απαιτεί εμπλοκή πολλών διαφορετικών εμπλεκομένων φορέων που πρέπει να καταλάβουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι διαφορετικοί επαγγελματικά. Πρέπει όμως να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που θα τους επιτρέπει να δουλεύουν με ασφάλεια, ισότητα και για την είσοδο και για τη σταδιοδομία και για την ανάπτυξη και να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα προσόντα και των ανδρών και των γυναικών. Είναι δυνατόν. Εγώ μπήκα σε, σε έφυξα ορισμένα ζητήματα. Είμαι έτοιμη να συζητήσουμε και γι' αυτό και για άλλα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, γύρατε διάφορα σημαντικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη το οικονομική μοντελοποίηση, πώς μπορούμε να εξετάσουμε τα διάφορα οικονομικά μοντέλα, ώστε να βρούμε απαντήσεις για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα θα σας δώσουμε την ευκαιρία να θέσετε ερωτήσεις ε, στις τρεις ομιλήτριές μας. Η κυρία Μπερισέλα από τη Ρουμανία είναι η πρώτη που θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Η Κυρία Πιτσέλ από την ε, Ρουμανία. I am Anna Burchel from Romania. Είμαι η Άννα Μπίρτσελ από τη Ρουμανία. Chambers of Romania. Thank you so much for... Σας ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή ημέρα της γυναίκας για αύριο στην Ρουμανία για να αντιμετωπιστεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στις ε, γυναίκες λάβαμε υπόψη μας ότι πρόσφατα η χώρα μας ότι η χώρα μας δεν ήταν ένα έθνος νοικοκυρών. Οι γυναίκες δηλαδή δεν είχαν ποτέ πρόβλημα να προσαρμοστούν στην ε, αγορά εργασίας. Το πρόβλημα ήταν τι γινόταν από τη στιγμή που άρχισαν να δουλεύουν. Μία πρόσφατη περίπτωση δείχνει αυτό το παράδειγμα τον καλύτερο δυνατό πρώτο, ε, τρόπο. Οι περικοπές των μισθών στο δημόσιο τομέα κατά 25% από την προηγούμενη κυβέρνηση ε, με επικεφαλή στον Εμίλ Μποκ ε, μείωσαν το δημοσιονομικό έλλειμμα στα πρώτα χρόνια της χρήση, αλλά αυτό έπληξε τι γυναίκες σε περισσότερο από τους άντρες, διότι οι γυναίκες ήταν ε, η πλειοψηφία ε, των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευση, όπου οι γυναίκες είναι ακόμα περισσότερες, οι μισθοί ήταν σημαντικά μικρότεροι από σε άλλους κλάδους. Η παρούσα κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει το κοινωνικό κλίμα με επαναφορά των μισθών στα επίπεδα πριν τι ε, ακόμα και αν αυτή η διαδικασία είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Η αγορά εργασίας όπως είναι σήμερα δείχνει μία ε, μεγάλη και αυξανόμενη έκθεση στον, ε, ε, των γυναικών στον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι γυναίκες γίνονται φτωχότερες, ε, ε απουσιάζουν όλο και περισσότερο από την εργασία και το εισόδημα και οι συντάξεις τους μειώνονται σημαντικά σε σχέση με τους άνδρες. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, έχω κάνει λάθος. Ε, στο πρώτο πάνελ έχουμε μόνο ε, σύντομε ερωτήσεις. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα φτάσω και σε ερωτήσεις. Απλά ήθελα να σας παρουσιάσω μια γενική εικόνα τη κατάσταση στη Ρουμανία. Θα ήθελα να, λοιπόν, να ρωτήσω το πάνελ, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει έναν πληθυσμό που γυράσκει. Να ζητήσω τη γνώμη σας λοιπόν για ποια μέτρα, τα τρία ας πούμε, ποια θα ήταν τα τρία καλύτερα μέτρα αντιμετώπισης των ε, προβλημάτων αυτών. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, θα έπρεπε να το είχα ήδη αναφέρει, ότι οι ερωτήσεις ε, στο πάνελ αυτό θα πρέπει να είναι σύντομες αρχικά. Επόμενος ε, ομιλητής, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξαιρετικέ παρουσιάσεις από τρεις εντελώ διαφορετικές οπτικέ γωνίες. Τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα του, ιδιαίτερα η αναφορά στο πώς θα πρέπει να εισαχθούν οι νέες δεξιότητες στις, ε, στην αγορά εργασία και στις ε, γυναίκες. Και το αυτό που εξάγω εγώ από όλη την ε, συζήτηση και τις παρουσιάσεις είναι ότι χρειαζόμαστε μια διαφορετική ψέγγιση και από την ε, ομιλία της ε, δεύτερης ε, καλεσμένης φάνηκε πόσο σημαντική είναι η πολιτική και η ανάμειξη των ίδιων των φορέων στην αντιμετώπιση της κρίσης. θα ήθελα πάρα πολύ να ζητήσω πληροφορίες από εσάς, ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Στην χώρα μου υπάρχει ε, έντονο το πρόβλημα ε, της ανεργίας στην ε, ομάδα των Ρωμά και γι' αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας, ιδιαίτερα επειδή αναφερθήκατε στις μετανάστριες. Εδώ στην Επιτροπή είχαμε ήδη τρεις εκθέσεις ε, σχετικές. Η τελευταία ήταν της κυρίας Μογάν Σαρτιέ που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Και είμαι σίγουρη ότι φέτος στην Επιτροπή αυτή θα ασχοληθούμε με παρόμοια ζητήματα και η εμπειρία σας λοιπόν θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος από τα Εθνικά Κοινοβούλια που θα ήθελε να πάρει το λόγο και να απευθυνθεί στους καλεσμένους. Παρακαλώ. Θα ήθελα να, να ρωτήσω τους καλεσμένους πώς θεωρούν ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι σημαντική. Ο πρωτογενής δηλαδή τομέας, πώς θα βοηθήσει στην απασχόληση των γυναικών στην Ευρώπη. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ε, χώρες υποένταξης, στις ε, χώρες που έχουν κάνει αίτηση. Στο παρελθόν ο τομέας αυτός απασχολούσε πάρα πολλούς εργαζομένους, ιδιαίτερα γυναίκες. Και εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίξει τις γυναίκες αυτές, θα έχουμε και έσοδα από την γεωργία. Θα βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με όπως είναι τώρα. Εσείς πώς ε, βλέπετε τον τομέα αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παρακαλώ. Μία τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις σημαντικές συνεισφορές σας για την σημαντική αυτή μέρα της γυναίκας. Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις, αρχίζοντας με το πώς βλέπετε την εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ισχύ, σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Και τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης ε, εκπροσώπησης των γυναικών στις θέσεις αυτές. Και επίσης, ε, πόσο βλέπετε τις ε, περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, και πώς νομίζετε ότι οι περικοπές αυτές επηρεάζουν τις γυναίκες και τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις αρνητικές αυτές επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεση και σε περίοδο που προσπαθούμε να μειώσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα. Η ανισότητα ανδρών και γυναικών σίγουρα είναι ένα, να υπάρχουν φαινόμενο και πώς οι χώρες που αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο την κατάσταση θα βελτιώσουν, θα συνεισφέρουν θετικά στην βελτίωση του επίπεδου ζωής. Με ποιες πολιτικές, τι προτείνετε εσείς. έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Επί πολλούς αιώνες οι άνδρες ήταν εκείνοι που είχαν τον τελευταίο λόγο στη λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, αλλά και άλλους τομείς πολιτικής. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το πρόβλημα αυτό, να το λύσουμε, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι άντρες βρίσκονται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων. Πιστεύετε πως είναι πολύ αργά για να αλλάξει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε τώρα στους ε, πανελίστες. Θα θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Παρακαλώ, αρχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας. Πιστεύω πως δύο ζητήματα προκύπτουν από αυτό. Είτε πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ισότητα των φύλων ξεχωριστά και καθ' είτε επειδή η ισότητα των φύλων είναι καλή για όλα τα υπόλοιπα, για όλους τους υπόλοιπους τομείς. Και πιστεύω πως ε, όλες αυτές οι ερωτήσεις σας έχουν καταδείξει την διαφορά και τις εντάσεις που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της εγείρανσης του πληθυσμού, διότι χρειαζόμαστε τις γυναίκες να δουλεύουν, να δουλεύουν για πολύ καιρό έτσι ώστε να συνεισφέρουν στις συντάξεις, να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Επίσης, η γεωργία είναι πολύ σημαντικός ε, παράγοντας. Το τελευταίο τώρα ερώτημα, δηλαδή το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανισότητα των φίλων Αυτό φαίνεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται καθαρά. Και όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται περισσότερη εκπροσώπηση των γυναικών στις ε, υψηλόβαθμες ε, θέσεις, ε, στις θέσεις εργασίας, στην λήψη αποφάσεων, στον οικονομικό τομέα. Και πιστεύω ότι δεν είναι επαρκές να είναι εθελοντικοί η μέθοδος ε, αυτή συμπερίληψης των γυναικών. Χρειάζεται ποσόστοση. Πρέπει να έχουμε μία άμεση ανταπόκριση στην αντιμετώπιση μας. Και ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε την καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στις ε, υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας είναι η εισαγωγή ποσοστώσεων. Ποσοστώσεων ε, εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων. Διότι χωρίς ποσοστώσεις και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των κυβερνήσεων δεν έχει αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών όσο θα θέλαμε. Να μιλήσω τώρα για το θέμα του γυράσκοντος πληθυσμού. Το έχουμε και αυτό στην Ιρλανδία. Πριν όμως μπω σε αυτό, έχουμε και άλλο πρόβλημα. Στην Ιρλανδία και αλλού, προφανώς. Πολλοί φεύγουν από τη χώρα, ψάχνοντας δουλειά αλλού. Στην Αυστραλία για παραδείγμα. Και αλλού. Οι Ιρλανδοί. Αλλά πρόκειται για μια μεγάλη ανησυχία για μια χώρα όπως την Ιρλανδία. Μίλησε κάποιος ε, για την γύρανση του πληθυσμού. Λάβετε υπόψη και το ότι πολλοί κόσμος φεύγει οδηγώντα την Ιρλανδία να χάσει ότι έχει επενδύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Και μιλάμε για άτομα που είναι απόφυτοι πανεπιστημίου. Προτείνω λοιπόν να επενδύσουμε όχι μόνο στην Ιρλανδία, παντού περισσότερο στην αύξηση του πληθυσμού, των νέων ιδίω. Επίσης να δούμε τι είναι ελκυστικό στους νέους. Τι εννοώ με αυτό. Να βάλουμε περισσότερα κονδύλια και πόρους στην υποστήριξη νέων, ιδίως με μεγάλα προσόντα, και να παράσχουμε καινοτόμε ιδέες. Θα μπορούσαμε επίση να δώσουμε ιδέες που θα βοηθούσαν τη δημιουργία των θέσεων εργασία. Σε ό,τι αφορά τη ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων, αν έχουμε μια ημερήσια διάταξη ισότητα στο τομέα της λήψη απόφαση, δεν θα έχουμε τεράστιες αποκλήσει όταν συζητούμε διαφορές μισθολογικές ή συνταξιοδοτικές. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και θα έπρεπε να το δούμε και αυτό το θέμα, όχι να μιλάμε μόνο. Θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε και το θέμα των ποσοστώσεων. Εμείς, αν μπορούσαμε να δούμε τον τρόπο κάλυψης του κενού της απόκλησης που υπάρχει στη, μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο λήψης αποφάσεων θα καλύπτουμε και άλλα σημαντικά θέματα. Να προσθέσω κι εγώ κάποια θέματα. Και σχόλια. Όντως, η γύρανση του πληθυσμού είναι θέμα. Υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορούν να γίνουν. Πρώτον, οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι υγιείς, άρα πρέπει να προωθούμε μοντέλα υγείας που δημιουργούν δράσεις προς όφελος όλων όταν χρειάζεται η κοινωνία περισσότερη κατάρτιση, περισσότερη ενημέρωση. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε την διαβίου μάθηση, ούτω ώστε να μπορεί κάποιος να αποκτήσει προσόντα μόνος του και να ανταποκρίνεται στις, αυξανόμενε αυξανόμενες απαιτήσει σε προσόντα της κοινωνίας κάθε φορά στη διάρκεια της ζωής του. Υπάρχουν οι έννοιες αλλά δεν είμαι βέβαιη κατά πόσον όλοι καταλαβαίνουν την ανάγκη συνεχούς ε, αύξησης των προσόντων. Το ότι υπάρχουν πολλοί ανεργοί δείχνει ότι αυτό δεν έχει καλυφθεί. Και αυτό πρέπει να είναι στην μέση διάταξη και των πολιτικών και των ηγετών που θα έπρεπε να προσπαθούν να βοηθήσουν, να διευκολύνουν αυτές τις δομές. Κάτι άλλο που σχολίασαν οι συνάδελφοι στο πάνελ έχει να κάνει με τη θέση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εγώ προσωπικά, για να σας πω την αλήθεια, είμαι αντίθετη με αυτό. Διότι στην ουσία το να δίνουμε προτεραιότητα στις γυναίκες αποτελεί μια διάκριση. Συμφωνώ μαζί σας ωστόσο ότι έχω αλλάξει, έχω τροποποιήσει την άποψή μου σχετικά. Όντως, πρέπει στο σύστημα λήψης αποφάσεων να υπάρξουν κάποιες αλλαγές που θα επιτρέπουν να καταλάβουμε ότι στην κοινότητα υπάρχουν γυναίκες ικανές που μπορεί να είναι στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση επιχειρήσεων. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η εισαγωγή ποσοστώσεων και έχουμε κάποια καλά παραδείγματα στην Ευρώπη, στη Σουηδία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία. Γίνεται σχετική συζήτηση στη Γερμανία και την Βρετανία. για πολλούς λόγους. Το θέμα εκεί είναι ποιος είναι ικανός, όχι αν άντρας ή γυναίκα. Δεύτερον, η δυναμική της διαχείρισης των επιχειρήσεων αλλάζει προς τη θετική κατεύθυνση. Και τρίτον, οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κρίσιμη κατάσταση ε, πιο οργανωμένα λόγω των φυσικών τους καθηκόντων. Επειδή πάντα είχαν πολλαπλές δουλειές, ήταν μητέρες, δούλευαν, είχαν το, το νοικοκυριό. Βέβαια, μη με θεωρήσετε ότι προσπαθώ να υποστηρίξω μια προνομίωχα θέση για τις γυναίκες, αλλά οι πολιτικές θα έπρεπε να παρέχουν τον καταλήτη το περιβάλλον, ένα περιβάλλον καταλήτη βάσει της αντικειμενικής πραγματικότητας. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, το θέμα είναι η ανάγκη νέας ανταγωνιστικότητας, το να βοηθήσουμε την Ευρώπη σήμερα μέσω και μακροπρόθεσμα. Δεν έχει να κάνει με την κατάσταση, την ατομική κατάσταση του Α ή του Β. Η τελευταία ερώτηση αφορούσε αποφάσεις που λαμβάνονται σε έτσι ανδροκεντρικό πλαίσιο. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να το προσεγγίσουμε διαφορετικά. Οι η υπεύθυνοι λήψη απόφαση σήμερα χρειάζονται για να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρώπη. Το θέμα της ισότητας είναι θέμα που επιτρέπει να υλοποιήσουμε ενεργά προγράμματα και να κάνουμε δραστηριότητες σε κάθε επίπεδο, σε εθνικό, σε τοπικό, σε επαγγελματικό και ταυτόχρονα διευκολύνοντας το περιβάλλον στην κοινότητα, παρέχοντας και προγράμματα για την υπέρβαση των ε, προκαταλήψεων και των στερεότυπων ήδη σε πολύ μικρή κατάσταση, διότι ο σημερινός δεκάχρονος και η σημερινή δεκάχρονη θα είναι αύριο τα αφεντικά στην κοινότητά μας. Χρειάζεται λοιπόν να δουλέψουμε με τα παιδιά και τις οικογένειες ώστε να αρχίσει να αλλάζει κάπως αυτή η νοοτροπία και να εισάγουμε νέα μοντέλα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ τις τρεις, ε, τα τρία μέλη του πάνελ που ήρθαν ε, σήμερα για να συμβάλλουν στο διάλογο αυτό και να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Σας ευχαριστούμε. And we, and we will now swap the panelists, so we're going to the panel. Θα αλλάξουμε πάνελ τώρα, περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Bien, euh, Προτείνω να αρχίσουμε ε, το δεύτερο τμήμα της ε, συζήτησής μας με το δεύτερο πάνελ. Λέγομαι Μογάν Σαχτιέ και είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών και ισότητα των Δύο Φύλων. Θα ήθελα να σας πω ότι Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι εδώ στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλω να το τονίσω. Είμαστε περήφανοι που προεδρεύει άντρα στην Επιτροπή Γυναικών. Διότι είμαστε καθόλου πεπισμένοι πως ε, η ισότητα των γυναικών στο χώρο εργασίας ε, είναι κάτι που θα κερδίσουμε αν ε, αναλάβουν αντίστοιχη δέσμευση και οι άντρες. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Γκούσταυσον καθώς ε, και όλους τους άντρες ε, που ήρθαν στη σημερινή συνεδρία. Δεν πρόκειται για έναν φεμινιστικό αγώνα, Όλοι μαζί από κοινού ε, θα οικοδομήσουμε με νέα πραγματικότητα που θα εξασφαλίζει την ισότητα των δύο φύλων. Αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό είναι το θέμα συζήτησης που μας απασχολήσει σε αυτό το πάνελ. Ανταλλαγή εμπειριών και βελτίστων πρακτικών από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχουμε τρεις ε, παρεμβάσεις. Σας παρακαλώ και απευθύνομαι στα μέλη του πάνελ να τηρήσετε αυστηρά το χρόνο αγόρευσης ε, ε, με τρόπο ώστε να έχουμε χρόνο στη συνέχεια για τις ερωταπαντήσεις. Η Βαρόνη Ντέτα Οκάθιν, που είναι πρόεδρος ε, της Υποεπιτροπής Εσωτερικής Αγοράς Υποδομών και Απασχόληση στη Βουλή των Λόρδων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το, η πρώτη ομιλήτρια. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε, που ήρθατε στο σημερινό μας ε, σεμινάριο κατόπιν δεύτερη μαρτυρία από την Ισπανία. Κάρμεν Κιντανίλια Μπάρμπα, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας του Κοινοβουλίου της Ισπανίας. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Και στα πλαίσια τη πάλι του ίδιου πάνελ. Ε, προσκαλώ τον ε, Ρούλαν Κάρτο, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ισότητα των Δύο φίλων ε, και Δικαιωμάτων των Γυναικών, γερουσιαστή. Είσαι Γάλλος, θα πάρει τρίτος το λόγο και χαιρόμαστε που θα κλείσει το πάνελ ένας άντρα. Θα ακούσουμε μαρτυρίες λοιπόν, αρχίζοντας με την Βρετανική εμπειρία. Έχετε 10 λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε και να συμβάλλω κι εγώ σε αυτή την τόσο χρήσιμη ε, εκδήλωση. Όπω είπατε, είμαι πρόεδρο τη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά στη Βουλή των Λόρδων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εντολή που έχουμε στην υποεπιτροπή μα, διότι ασχολούμαστε με τι ε, υποδομέ Επιτροπή Εσωτερική Αγορά ε, και Απασχόληση. Ε, βέβαια, αυτά τα λέω γιατί είμαι πρόεδρο τη υποεπιτροπή. Α κοιτάξουμε λοιπόν από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία την εντολή που έχει λάβει η Επιτροπή μας. Ε, δεν αληθεύει ότι ασχολούμαστε μόνο με τα βρετανικά ζητήματα. Εξετάζουμε όλες τις οδηγίες, τα σχέδια, τη ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισμένες φορές ζητάμε έρευνες για την εκπόνηση εκθέσεων και τη συλλογή ε, τεκμηρίων. Ε, θα ήθελα σήμερα να εξετάσουμε όλος ιδιαιτέρως με ποιο τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι ούτως ώστε να εκπροσωπούνται καλύτερα οι γυναίκες σε υψηλό στο χώρο εργασίας. Για ποιο λόγο, διότι οι νέες γενιές, η νέα γενιά γυναικών καλύτερα καταρτισμένων, με καλύτερες ευκαιρίες να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια, ε, είναι ε, πολύ καλά επιμορφωμένες, όπως λένε στη ΣΑΒΙ, όπως λένε στη ΣΥΠΑ, ε, και έχουν τα προσόντα στη διάθεσή τους για έναν αυξημένο ρόλο στο χώρο εργασίας. Έχουμε κοινή ευθύνη όλοι μας ε, για να ενθαρρύνουμε τη νέα γενιά, όχι να κοιτάζουμε πίσω την ύφεση και όλα τα προβλήματα, αλλά να έχουμε μια μελλοντοστραφή προσέγγιση. Η Επιτροπή μας εκπώνησε μια έκθεση για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια μετά από μια έρευνα για την ισότητα των δύο φύλων ε, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ε, μας εξέπληξε ο χαμηλός αριθμός γυναικών σε θέσεις όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω έχουμε σημειώσει πρόοδο και δεν μα αναγνωρίζεται πάντοτε. Το 94 παραδείγματο χάρη, όταν διορίστηκα ε, πρώτη, πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο μια επιχείρηση ε, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ήμουν μία από τι έξι γυναίκε ε, που δούλευαν σε αυτή την επιχείρηση και τότε ήταν 1.800 οι γυναίκες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δηλαδή το ποσοστό των γυναικών ήταν 0,3% και 99,6% ήταν άντρε. Τώρα με τα νέα στοιχεία και την έκθεση από το Επαγγελματικό Φόρουμ των Διοικητικών Συμβουλίων μας ε, έδωσε στοιχεία βάσει των οποίων ε, αντί για 6 γυναίκες στο διοικητικά συμβούλια έχουμε 315. Δηλαδή, ε, ένα τέταρτο των διοικητικών συμβούλων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων έχουν εκπληρώσει το στόχο του 25% γυναικείας εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια. Ξέρω ότι έχει περάσει χρόνος από το 1994, είναι μεγάλο άλμα, μεγάλη πρόοδος. Και μόνο 7 επιχειρήσεις ε, του ΦΟΥΣ 100 είναι αποκλειστικά αντρικές επιχειρήσεις ε, σε εισαγωγικά. Τώρα όμως δακτυλοδεικτούνται από όλους και άρα μπορούμε να πούμε ότι είχαμε μια θετική επίπτωση με τη δράση μας ε, και ξέρω ότι οι ποσοστώσεις δεν είναι ε, πανάκια. Ε, εξάλλου αυτά τα καταφέραμε χωρίς ποσοστώσεις, απλώς όλοι ανέλαβαν το ρόλο και λειτουργήσαν υποδειγματικά αν θέλετε. Ε, τώρα, χωρίς ε, να γινόμαστε, γινόμαστε δογματικοί, θα δούμε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το 45% στην αγορά εργασίας είναι γυναίκες ε, και το 60% των αποφύτων είναι γυναίκες. Αλλά δεν επαρκεί κατά τη γνώμη μου αυτό. 17,3% μόνο στα διοικητικά συμβούλια στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι γυναίκες. Ε, το Πανεπιστήμιο Κανεφίλ επιβεβαίωσε σε μία έκθεση ότι οι γυναίκες που δύναται να, να αναλάβουν τέτοιες υψηλόβεθμες θέσεις έκανε μία έρευνα και έδειξε ότι υπάρχουν 500 γυναίκες οι οποίες γεννιούνται έτοιμες λόγω εκπαίδευσης ε, και ε, καταγωγής. Ε, αντίστοιχα δεδομένα υπάρχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα στοιχεία που συλλέξαμε διαπιστώσαμε ότι η κοινωνία και οι επιχειρήσεις θα υποφεληθούν τα μαλά από την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Φυσικά είναι δύσκολο να το αποδείξουμε αυτό, να συνδέσουμε τα κέρδη μιας επιχείρησης με τα αυξημένη συμμετοχή των γυναικών, όμως αποδείξαμε ότι ε, με μια αυξημένη συμμετοχή ταλαντούχες γυναίκες θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας ε, και έτσι θα έχουμε ένα ευρύτερο φάσμα ιδεών αποφεύγοντας το groupthink το υπονομαζόμενο επικεντρωμένο δηλαδή ε, στις αντρικέ εισαγωγικά ιδέε. Λοιπόν, για τα διοικητικά συμβούλια στις επιχειρήσεις είδαμε επίσης ότι Αυτά τα στοιχεία μπορούν να μας βοηθήσουν ε, για να ε, πραγματευτούμε το ε, θέμα συζήτησης του σημερινού πάνελ. Ε, ε, με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν θετικά παραδείγματα βελτίστων πρακτικών από πλευρά των εθνικών κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι πολλέ χώρε, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ενσωματώσει έμφυλε απαιτήσει στο εταιρικό του δίκαιο. Παραδείγματο χάρη, το εταιρικό δίκαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, προτάσει τη σημασία τη ε, διαφορετικότητα ω προ την κάλυψη υψηλόβαθμου θέσεων στα ε, διοικητικά συμβούλια και υπάρχει και μια επιτροπή διορισμών όπου εκπονούνται προδιαγραφέ σε σχέση με την έμφυλη κατανομή των θέσεων και την εκπλήρωση των έμφυλων στόχων από πλευρά των επιχειρήσεων. Βάσει ετησίων εκθέσεων για τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια υποχρεούνται οι αρμόδιοι να συνυπολογίσουν αυτό τον παράγοντα της ε, ε, ε, ίση συμμετοχή των ανδρών και γυναικών. Βεβαίως με την πολιτική λιτότητα και την ύφεση βλέπουμε ότι υποχωρεί η θέση των γυναικών δυστυχώς στα διοικητικά συμβούλια όλοι μας ε, έχουμε κάποια ευθύνη και στον πολιτικό βίο αλλά και στον επιχειρηματικό βίο να προσπαθήσουμε ε, να μειώσουμε αυτή, αυτή την αίσθηση απόγνωσης ε, που αποτυπώνεται στα μυαλά των νέων γυναικών λόγω της κρίσης. Βλέποντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ειχέγγυα για τους νέους ε, που θα μετουσιωθεί σε ένα σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων προς τα κράτη-μέλη ώστε να προσφέρουν σε απασχόληση στις γυναίκες ε, βλέπουμε ότι τέσσερις μήνες ε, μετά την αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο εμ, εμ, καταγράφονται ως άνεργες πολλές γυναίκες και αυτό είναι λυπηρό. Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο για να δώσουμε μια απάντηση στην κρίση τις ανεργίες και να γνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κέριο ρόλο για να προσδώσει νέα κίνητρα στις ε, κυβερνήσεις, ε, να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βελτίωση των πρακτικών ανάμεσα στις κυβερνήσεις και είδαμε πολύ παραδείγματα σήμερα το πρωί και ε, θα διαβιβάσω όλα αυτά τα στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να εργαστούν σε τέτοιες επιχειρήσεις, υπάρχουν και άλλα σοβαρότατα προβλήματα για τις γυναίκες. Παραδείγματο χάρη, μία πρόσφατη έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο Βασίλειο είδαμε ότι οι περικοπές στο δημόσιο τομέα έπληξαν ιδιαίτερω ε, τι ε, γυναίκες. Τα ακούσαμε εξάλλου αυτό σήμερα το πρωί περίπου 40% ε, των θέσεων απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο των γυναικών ε, είναι στο δημόσιο τομέα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι περικοπές στο δημόσιο τομέα ε, θα έχουν δυσανάλογα μεγάλο αρνητικό αποτέλεσμα για αυτέ τι γυναίκες. Σε βάση τη ίδια έρευνα είδαμε ότι οι γυναίκες δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε καλέ θέσει εργασία και σε περίθαλψη για τα παιδιά του σε προσιτέ τιμές και έτσι συνδέονται με το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών με τις επιπτώσεις της τωρινής ε, κρίσης ε, και ε, θα ήθελα να αποκομίσω περισσότερα στατιστικά στοιχεία για αυτό το ζήτημα από τη σημερινή μας συζήτηση. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να μην προ... εστιάζουμε τόσο πολύ στα προβλήματα διότι είναι βρέχη πρόθεσμα και αλλάζουν τα δεδομένα καθημερινά. Δείτε τι γίνεται στα χρηματιστήρια καθημερινά. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι ε, ε, όχι τόσο το παρελθόν. Λέμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, παράλυση by Άμα τα παραναλύουμε τα πράγματα, παραλύουμε και δεν κάνουμε τίποτα. Α σταματήσουμε λοιπόν να ασχολούμαστε ε, με ε, θεωρητικά με τις επιπτώσεις ε, της κρίσης ε, ε, και να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε νέες δράσεις όπως είδαμε από αυτή την λαμπρή εκπρόσωπο της Hewlett Packard που δεν είναι και η μόνη παραδείγματος χάρη στην κοινωνία της πληροφορίας υπάρχουν πολλές νέες θέσεις απασχόληση εξ αποστάσεως κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντικό ας μην ασχολούμαστε με το παρελθόν ε, γιατί φθήνουν αυτές οι παλιές βιομηχανίες. Ας κοιτάξουμε προς το μέλλον και ας δούμε ποιοι θα είναι οι πλέον ανταγωνιστικοί τομείς στο μέλλον ε, και να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τη μεταποιητική βιομηχανία που παρατηρούνται και οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης για τις γυναίκες. Λοιπόν, ε, να μία βιομηχανία που πνέει τα λίστια και βλέπουμε συγκεκριμένα στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι φθήνει αυτή η βιομηχανία και ανθούν καινούργιες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία που μας δώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά περιόριστε σας ευχαριστούμε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να έχουμε την ανάλυση και την ε, πεφωτισμένη παρουσίασή σας. Περνάμε τώρα στην Ισπανία. Έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά κι εσείς. Και κατόπιν θα μιλήσουμε την παρέμβασή σας. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτον, θα ήθελα να σας καλημερίσω όλους σας κυρίες και κύριοι και να ευχαριστήσω την Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, ευγενική της πρόσκληση που μου επέτρεψε να έρθω εδώ και που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρε της Ένωσης, ιδίως δε οι γυναίκες. Οι γυναίκες σε μια εποχή οικονομικών δυσκολιών, όπου όπως σωστά αναφέρει το πάνελ, η υπέρβαση της κρίσης και οι βέλτιστες πρακτικές των, Εθνικών Κοινοβουλίων. Και εγώ αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσω για το Εθνικό Κοινοβούλιο της Ισπανίας. Θέλω επίση να σας πω ότι έχω μαζί μου την Αντιπρόεδρο της ε, Επιτροπής, κυρία Τρινιδάδ Χιμένεθ, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και, πρόεδρο, και την Πρόεδρο της Επιτροπής Όντας της Ισπανικής Γερουσίας, κυρία Κάρμεν Τράις. Έχουμε λοιπόν παρουσία εδώ η Ισπανία για να μιλήσουμε για το πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει τις Ισπανίδες. Περνάμε μία από τις πιο σκληρές στιγμές ε, της σύγχρονης ιστορίας όλων των χωρών της Ένωσης. Πολύ σωστά το είπε ο αντιπρόεδρος κύριος Πιτέλα, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Έχουμε μία κρίση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αν δεν θέλουμε να φέρουμε στο μυαλό μας την μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 20 Σήμερα στον 21ο αιώνα πρέπει να δούμε τι μέλλον θα δώσουμε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για να βγάλουμε εκατομμύρια ανθρώπων από μια θλιβερή οικονομική κατάσταση. Βεβαίως η Ισπανία δεν είναι μια απομονωμένη κατάσταση, βιώνει με σκληρό και έντονο τρόπο την οικονομική κρίση. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Ισπανίας αντιμετωπίζει αυτή την οικονομική κρίση με μεταρρυθμίσεις που παρουσιάσαμε στην Ένωση για τον τρόπο με τον οποίο μειώσαμε το έλλειμμα και το δημόσιο ε, χρέος, ε, το έλλειμμα της χώρας από το 9,1% στο 6%. Αυτό μας επιτρέπει να ανοίξουμε μία πόρτα ευκαιρία και να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να γυρίσουμε, να πιστέψουμε στην ανάπτυξη, στην, ε, οικονομική, ε, στην οικονομική ανάπτυξη, στην ανάκαμψη και, στην, ε, και το πόσο καθένας μπορέσει να μας επιτρέψει να, να μας, και το πόσο το κάθε, η κάθε εξέλιξη αυτή θα μας βοηθήσει. Αλλά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην Ισπανία, τα στοιχεία της ανεργίας ε, δείχνουν ότι η κρίση επηρέασε σημαντικότερα τον κλάδο της κατασκευής, τον κατασκευαστικό τομέα. Είναι προφανές. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ο αριθμός των ανέργων, ανδρών ή γυναικών, είναι ίδιος. 2,5 εκατομμύρια είναι οι γυναίκες, 2.507.000 ε, είναι οι γυναίκες, 2.482.000 οι άνδρες. Τα στοιχεία των ατόμων που δεν έχουν εργασία άνω των 25 είναι αντίστοιχα. 2.150.000 γυναίκες, 2.226.980 άνδρες. Γιατί μιλάμε λοιπόν σήμερα. Για το πώς επηρεάζει η κρίση τους άνδρες και τις γυναίκες. Για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη συζήτηση για την ισότητα εμπλέκοντας αναγκαστικά τους άνδρες στην πρόοδο των γυναικών και στις δεμεύσεις για την ισότητα των φύλων για να μπορέσουμε να δούμε το πώς θα φτιάξουμε έναν πιο δίκαιο κόσμο. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι σήμερα η οικονομική κρίση οδηγεί περισσότερες γυναίκες στη φτώχεια. Η οικονομική κρίση σήμερα γυρίζει τις γυναίκες που χάνουν τη δουλειά τους στο σπίτι τους και χρειάζονται να κάνουν, να αναλάβουν τον οικοκυριό τους, όχι μόνο με λιγότερους πόρους, αλλά και με μικρότερη ελευθερία, να αναλάβουν επιπλέον την ε, φροντίδα των παιδιών και των γονέων με ακόμα μικρότερο, με ακόμα μικρότερη αγοραστική ε, δυνατότητα. Το θέμα το είχαμε αντιμετωπίσει στην Ισπανία σε πολλές ε, και με διάφορες κοινοβουλευτικέ πρωτοβουλίες, τόσο στην ισότητα, στην Επιτροπή ισότητα του, του, του βουλή της Βουλής, όσο και της Γερουσίας. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε στενή συνεργασία με τις ε, δομές ε, εκπροσώπησης των γυναικών. Είδαμε την κατάσταση ζητώντας την υιοθέτηση μέτρων που θα επιτρέπουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας για γυναίκες άνω των 45, ε, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για γυναίκες κάτω των 25. Την κρίση την ε, είδαμε και από το ξεκίνημα μιας συζήτησης όπως τέθηκε και στο προηγούμενο, στο προηγούμενο πάνελ την ε, μισθολογική διαφορά που επηρεάζει την ε, ζωή των γυναικών. Μία κατάσταση που ε, αυτό το κενό είναι 16,5% στην Ισπανία. Ο μέσος όρος των 25 χωρών της Ένωσης που είναι 16,4%. Επιπλέον, η, ανισο, η μισθολογική ανισότητα οφείλεται εν πολλής και στο στην, στις ώρες δουλειά των γυναικών. Το 73% των, γυναικών, των ατόμων που δουλεύουν με μερική απασχόληση στην Ισπανία είναι γυναίκες. Εξού και, και εκεί ακόμα η διαφορά, η μισολογική διαφορά των γυναικών είναι 8, περισσότερο 8% περισσότερο για τις γυναίκες στην, στις συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε σχέση με όσους ε, δουλεύουν πλήρη απασχόληση. Από την άποψη αυτή, οι διάφορες, ε, τα διάφορα κόμματα στην Βουλή και την Κυρισία από κοινού ζήτησαν από την κυβέρνηση να προωθήσει τη μισολογική ισότητα με ένα πιο ισχυρό και έντονο μοντέλο στρατηγικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που περιλαμβάνονται στη στρατηγική 2015 της Επιτροπής. Ζητήθηκε επίσης από την πρωτοβουλία αυτή να ξεκινήσουν μέτρα που θα επιτρέπουν την ισότητα, τη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια δουλειά ή για αντίστοιχη αξίας δουλειά. Ζητήσαμε επίσης την εφαρμογή του άρθρου 45 του νόμου για την, ισότητα, την αποτελεσματική ισότητα ευκαιριών ένα νόμο του 2007 να υλοποιηθεί πραγματικά η μάχη κατά της μισθολογικής ανισότητας. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η αρχή, η Επιτροπή Ισότητας των Κοινοβουλίων και του Ισπανικού Κοινοβουλίου ε, παροτρύνει με αποτελεσματικό και σαφή τρόπο μέτρα για την υλοποίηση δεσμεύσεων πρόσβαση στην αγορά εργασίας και μείωση της ε, μισθολογικής ανισότητας, ζητώντας από την κυβέρνηση να προβεί σε μια ουσιαστική και πραγματική διάγνωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας όπου δουλεύουμε με αποφασιστικό και ειδικό τρόπο. Να σας πω επίσης ότι η δουλειά που κάνει η Επιτροπή Ισότητας ε, στο Ισπανικό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντική. Σήμερα, ε, σε μια εξαιρετικά σκληρή κρίση, όταν κάθε μήνα βλέπουμε πώς χάνονται θέσεις εργασίας, πώς δυστυχώς αυτή η οικονομική κρίση επηρεάζει με εξαιρετικά σκληρό τρόπο τις γυναίκες και το πρόσωπο των γυναικών στον κόσμο είναι το πρόσωπο της φτώχειας, όταν η ισότητα σημαίνει και το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δουλεύουμε για την απασχόληση, για να σπάσουμε τη διάκριση που υφίστανται οι γυναίκες, ξεκινήσαμε στην Επιτροπή Ισότητας, Επιτροπή, για να μελετήσει τον εξορθολογισμό των ωραρίων και την συνδιαλλαγή επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής καθώς και τη συνυπευθυνότητα ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, ένα κρεμές θέμα σε πολλές χώρες της Ένωσης, αλλά αναδιαμφισβήτητα και στην Ισπανία. Μου λένε ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι όταν μιλάμε για νομοθετικές πρωτοβουλίες, μιλάμε και για το τι κάνει η κυβέρνηση της Ισπανίας η κυβέρνηση της Ισπανίας μαζί με τις κυβερνήσεις των αυτονόμων κοινοτήτων περιφερειών υλοποιεί μέτρα που επιτρέπουν την πρόσληψη ανδρών και γυναικών με μίνιμουμ περίοδο 6 μηνών και επιδότηση, ενίσχυση πιο σωστά, 2.700 ευρώ για περίπτωση γυναίκας και 2.400 ευρώ για περίπτωση ανδρών. Για τους νέους μιλώ γιατί πρέπει να χτυπήσουμε την ανεργία των νέων και την ανεργία που πλήττει εκατομμύρια γυναίκες και εκατομμύρια άντρες. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει νομοθετικό έργο, τι σημαίνει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία σε αυτό το έργο δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η προηγούμενη ομιλήτρια, η, η Βαρόνια Κατάιν, είπε κάτι σημαντικό. Πρέπει να πάψει η ψύχωση της οικονομικής κρίσης που ε, κυριαρχεί σε εκατομμύρια άτομα στην Ένωση. Η κρίση δεν πρέπει να οδηγήσει στην κατάθλιψη εκατομμύρια άτομα. Γι' αυτό είναι σημαντικό ως κοινοβούλια, ως βουλευτές να προχωρήσουμε με έναν παιδαγωγικό τρόπο. Να δείξουμε ότι μπορούμε με θυσίες και προσπάθειες να βγούμε από αυτήν την τόσο σκληρή και, δυστυχώ, και, και θλιβερή κατάσταση που βιώνουμε σε πολλές χώρες στην Ένωση. Την οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Κλείνω λέγοντας σας κάτι σημαντικό. Εγώ γύρισα από τη Νέα Υόρκη. Μετέσχον εκεί σε μια συνάντηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα Περισσότερο από ποτέ πρέπει να προχωρήσουμε μαζί. Η Ένωση δούλεψε, δουλεύει από κοινού στο πλαίσιο της Ένωσης. Όταν δουλέψουμε για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις του Πεκίνου, τις τέταρτης, τις διεθνούς διάσκεψης του, του Πεκίνου, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση για το, την ισότητα στο μέλλον ανδρών και γυναικών. Πέρυσι δεν βγήκε το τελικό κείμενο. Πέρυσι η... το πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών ήταν ε, γυναίκες στη δουλειά. Δεν βγήκε το κείμενο εκείνο. Τώρα δουλεύουμε για το φετινό κείμενο. Βία, έμφυλη βία. Η βία που υφίστανται εκατομμύρια γυναίκες στο, στο στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει ενιαία Υπάρχει ωστόσο κάποια χώρα που δεν διαπραγματεύεται. Υπάρχουν χώρε που δεν διαπραγματεύονται με την Ένωση. Πρέπει να προχωρήσουμε μαζί για να δημιουργήσουμε το μέλλον εκατομμυρίων γυναικών στον κόσμο. Ζήτω συγγνώμη διότι ξεπέρασα τον χρόνο. Ευχαριστώ. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, τρίτη μαρτυρία. Πρόεδρος ε, Γολάν Κουχτό, ε, θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε τις ε, γαλλικές πολιτικές στους κόλπους της Γερουσίας για το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 100% συμφωνώ με τα, τις παρατηρήσεις που ακούσαμε από την προαλή σας. Το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών δεν είναι ζήτημα των γυναικών αποκλειστικά. Ακούστηκε ήδη αυτό σήμερα στη συζήτηση και μεταξύ άλλων ένα από τους λόγους για τους οποίους ήρθα εδώ για να εκπροσωπήσω τη γαλλική γερουσία. Ε, μετά τις επιπτώσεις ε, της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη και τον κόσμο ε, θα πρέπει να η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να εμπλακούν σε αυτόν τον κοινό καθημερινό αγώνα υπεράσπισης της απασχόλησης και προστασίας ε, των συμπολιτών μας, ε, γυναικών και αντρών, ε, από την κρίση. Χρειαζόμαστε πολιτικές και πρέπει να εμπνευστούμε από τους εταίρους και τις γειτονικές μας χώρες. Γι' αυτό είναι πνόμο προς την Επιτροπή των Γυναικών και Ισότητας των Δύο Φίλων και όλος ιδιαίτερος προς τον πρόεδρο Μάικλ Γκούσταυσον, χάρη στην πρωτοβουλία του οποίου συνεδριάζουμε σήμερα για να εξετάσουμε αυτό αυτό το ζήτημα. Ποιος είναι ο ρόλος των γυναικών λοιπόν ε, Ποιο μπορεί να είναι ο ρόλο των γυναικών για να μετριαστούν τα αποτελέσματα της κρίση και να βρούμε κάποιε απαντήσει. Ε, Θα ήθελα να σα παρουσιάσω τι νομοθετικέ ε, διατάξει που συζήτησε και ενέκρινε το Γαλλικό Κοινοβούλιο και τα δύο σώματά του, καθώ και τι συστάσει που εκπώνησε η Αντιπροσωπεία των Δικαιωμάτων των Γυναικών της Γερουσία, συμβάλλοντα έτσι στο τρέχον πρόγραμμα της γαλλικής κυβέρνησης. Θα ήθελα να τονίσω όλος ιδιαίτερους τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης ε, των δύο φύλων και σήμερα πλέον δεν θεωρείται ότι είναι μια απέτηση για να επικρατήσει κοινωνική ισότητα, θεωρείται μοχλός ε, για να βελτιωθεί η ποιότητα της ε, διαχειριστικής πολιτικής των επιχειρήσεων και όχι μόνο, αλλά και των κρατών μελών. Εδώ και χρόνια έχουν γίνει μελέτες στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ που έδειξαν ναι, ότι η, ισότιμη, η πιο ισότιμη εκπρόσωπηση των δύο φύλων ε, συνιστά ένα σημαντικό ατού ε, για τις επιχειρήσεις διότι προτείνει ένα διαφορετικό διαχειριστικό στυλ ε, στις επιχειρήσεις και οι γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι προφανές ότι η αυξημένη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων δεν είναι αυτή καθ' αυτή πανάκια, όμως ας μην υποτιμάται η σημασία της σε περίοδο κρίσης. Η Γαλλία σε αυτό το τομέα θέλησε να έχει ρόλο πρωτοπόρου και θέσπισε ποσοστώσεις που επιτρέπουν αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στα διευθυντικά διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων στη Γαλλία. Ε, οι Γάλλοι βουλευτές, ε, κυρίως ε, η Μαρίζο Ζίμερμαν που ήταν τότε πρόεδρος Επιτροπή Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών του Γαλλικού Κοινοβουλίου αγωνίστηκε σκληρά για αυτό το θέμα και τη αποτείω φόρο στις 27 Ιανουαρίου 2011 ενέκρινε το Γαλλικό Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο σε σχέση με τις ποσοστώσεις για τα διοικητικά συμβούλια των συγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και των δημοσίων επιχειρήσεων. Τρία χρόνια μετά τη θέση ισχύ του νόμου 2014 δηλαδή, τα εν λόγω συμβούλια θα πρέπει να έχουν 20% γυναίκες. Έχει ήδη εγκριθεί, είναι ένα κεκτημένο αυτό πλέον. Τρία χρόνια μετά το 2017 δηλαδή το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να ανέλθει στο 40%. Οι διατάξεις αυτές ε, ήδη έχουν οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Τον Οκτώβριο 2012 έγινε μια μελέτη που μας έδειξε ότι τα διοικητικά συμβούλια των 40 μεγαλύτερων γαλλικών επιχειρήσεων έχουν αυτή τη στιγμή ήδη δηλαδή 25% γυναίκες. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση επίσης ε, απεφανθεί για την, ε, το σχέδιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας για μια καλύτερη και πιο ισόρροπη συγγνώμη, εκπροσώπηση των γυναικών σε επίπεδο στελεχών στις επιχειρήσεις και το 2013 η Γαλλική η Γερουσία ε, προσυπέγραψε αυτό το στόχο του 40% για τη συμμετοχή των γυναικών στα συμβούλια. Πέριψε όμως ε, τα εκτελεστικά μέτρα για την πρόσληψη των διευθυντικών στελεχών καθώς και την δυνατότητα εξαιρέσεων που αποδυναμώνουν το σχέδιο οδηγίας αντίθετα. Επιθυμεί να υιοθετηθούν φιλόδοξοι και δεσμευτικοί ευρωπαϊκοί κανόνες και το τονίζω αυτό αυτό τέλος. Η Γαλλία έχει ένα μηχανισμό που εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο τομέα με την, το νόμο του, της Μαρτίου 2012. Σταδιακά θα εφαρμοστούν ποσοστώσεις για τις, ε, ε, ε τους ετήσιους διορισμούς σε διευθυντικές ε, σχέσεις, ε, ε, θέσεις συγγνώμη, στο δημόσιο τομέα. 60% των διορισμών από το Μάιο του 2012 μέχρι ε, σήμερα ήταν γυναίκες. Η πρόταση της κυβέρνησης ε, απορρέει από τον πρόεδρο της Δημοκρασίας, το ξέρετε, και από τον Πρωθυπουργό κοινοβούλιο λόγω ε, του διαχωρισμού των εξουσιών δεν έχει ε, τόσο ευρειε αρμοδιότητες. Όμως από το Μάιο του 2012 έχουμε ε, κυβέρνηση με ισότιμη, ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων για πρώτη φορά στην ιστορία. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη σημασία αυτού όταν εξετάζουμε το θέμα της ισότιμη εκπροσώπησης των γυναικών στις υψηλόβαθμέ θέσει και την που έχει αυτό για το στη διαχείριση σε επίπεδο κυβέρνηση και επιχειρήσεων. Η αρμόδια υπουργό επίση συνόδευσε αυτό το νομοσχέδιο με μέτρα που επιτρέπουν ε, να λαμβάνονται διαρκώ νέα μέτρα και εκτελεστικέ διατάξει μετά από την έγκριση αυτού του νομοσχεδίου, εξασφαλίζοντα έτσι ε, την ισότιμη εκπροσώπηση. Ε, καταπολεμούνται επίση τα στερεότυπα. Ξέρετε ότι με τους νέους νόμους επιταχύνονται οι εξελίξεις, αλλά χρειάζεται κάτι παραπάνω για να αλλάξουμε τις νοοτροπίες και πρέπει να αρχίσουμε τις προσπάθειες ήδη από, ε, τη, ε, από μικρές ηλικίε, ε, στα νήπια αγωγεία παραδείγματος χάρη, γιατί εκεί γεννώνται ε, τα στερεότυπα και τα κλίσε. Για να εξασφαλίσουμε την ισότητα των δύο φύλων, ε, το χρεια... δημιουργήθηκε μόλις τώρα το Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων από ε, τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει και το θέμα της βίας που ασκείται κατά ε, των γυναικών. Ε, αυτό είναι εκ των ουκ άνευ. Πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους μας σε αυτό το τομέα προτού κάνουμε οτιδήποτε άλλο και μάλιστα σύντομα εγκρίθηκε ένα σχετικό νομοσχέδιο για να παταχθεί η βία κατά των γυναικών. Εν γέννη θα πρέπει οι δημόσιες πολιτικές μας να συνυπολογίζουν την έμφυλη διάσταση ε, όλων των ζητημάτων, κυρίως για τις ευπαθέστερες κοινωνικές ε, ομάδες ε, που πλήττονται από την κρίση και αυτό είναι το δεύτερο τμήμα της παρέμβασής μου. Τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ξεκάθαρα ότι ε, οι γυναίκες που αντιστοιχούν στο ίμιση του ενεργού πληθυσμού ε, ε, αντιστοιχούν στο 75% των χαμηλών δεν έχουν εξίσου πολλές δεξιότητες όπως οι άντρες, ταυτόχρονα όμως καλύπτουν εκείνες τις βιοποριστικές υπηρεσίες όταν μιλάμε για τον τομέα των υπηρεσιών, για τα δίκτυα διανομής και γενικότερα καταλαμβάνουν ως επιτοπλίστων χαμηλόμιστες θέσεις εργασίας. Με την κρίση λοιπόν θα βουλιάξουν ακόμη περισσότερο στη φτώχεια, την ύφεση και θα καταστεί ε, επισφαλέστερη η θέση τους. Ε, στη συνέχεια καταργούνται ε, μαζικά θέσεις απασχόλησης σε κατεξοχήν αντρικό ε, σε εισαγωγικά οικονομικούς ε, τομείς ε, φαίνεται ότι ο τομέας των υπηρεσιών δεν έχει πληγεί τόσο πολύ. Όμως το 2009 άρχισε να αυξάνεται η ανεργία των γυναικών και το 55% των ανέργων είναι γυναίκες πλέον. Οι γυναίκες δεν υποαπασχολούνται διότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται μερικών αλλά και η ίδια η μερική απασχόληση έχει ε, περισταλεί και έχει φτάσει στις 15 ώρες εβδομαδιαίως. 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι πλήττονται από αυτά τα δεδομένα χαμηλών δεξιοτήτων είναι και το ποσοστό των γυναικών είναι 85% και παραμένουν έγκλειστες σε αυτή την επισφαλή θέση και σε αυτή την φτώχεια και την ύφεση. Ε, ε, θεσπίζονται διάφορες νέες εγγυήσεις από την κυβέρνηση, όμως ε, υπάρχουν δυνατότητες εξαίρεσης σε σχέση με τις συλλογικέ συμβάσεις. Η μερική απασχόληση σημαίνει χαμηλόμιστες θέσεις απασχόλησης με κειμενόμενα ωράρια, μειωμένη πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και όπως σας είπα η μερική απασχόληση έχει ήδη παρουσιάσει μείωση ως προς τις ώρες εργασίας εβδομαδίως. Ε, θα κλείσω, Πρόεδρε, η αντιπροσωπεία μας ε, στην Γερουσία ε, έχει εκδώσει μία σειρά συστάσεων το 2011 σε σχέση με τις ώρες εργασίας, σε σχέση με την προθεσμία προειδοποίησης για απόλυση, για καλύτερη πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες και τέλος το κράτος αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι και θα κλείσω έχουν από κοινού ε, κατευθυνθεί προς μία εθνική συμφωνία που στις 11 Ιανουαρίου 2013 υπεγράφηκε και προβλέπει μία μισθολογική άξιση για τις ε, υπερορίες καθώς και μία ελάχιστη διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας ε, που έχει οριστεί στις 24 ώρες την εβδομάδα. Αυτό ισχύει και για τους φοιτητές ε, κάτω από τον 25, όχι μόνο για τις γυναίκες. Όλα αυτά τα μέτρα θα εγγραφούν στο εργατικό δίκαιο με ένα σχέδιο ένα νομοσχέδιο που τώρα εξετάζεται από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Για αυτή την μαρτυρική σας κατάθεση. Οχτώ άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Μαρτυρίες από διάφορες ε, κοινοβουλευτικούς. Θα ζητούσα να τηρήσετε αυστηρά το δίλεπτο παρέμβασης για να προλάβουμε την καθυστέρησή μας. Δίνω το λόγο στην κυρία Ματράη από την Ουγγαρία ορμόμενη. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Πρόεδρε, η ασφάλεια, η οικογενειακή ασφάλεια σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι πολύ σημαντική, έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να συνδυάσουν εργασία και οικογένεια. Στην στρατηγική 2020 αυτό πώς ε, φαίνεται, με προγράμματα μεταρρυθμιστικά τα οποία πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη, τα οποία θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα, όπως για παράδειγμα το ε, χρέος, το οποίο πλήττει κατά κύριο λόγο τους ιδιώτες. Και έγινε ορατό από το 2009 το πρόβλημα αυτό. Από τότε βέβαια μέχρι τώρα έχει αυξηθεί δραματικά, έχει αυξηθεί επίσης δραματικά και το ποσοστό της ανεργίας. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προσπάθησε μέσω της απασχόλησης και μέσω της ε, φορολογίας να δημιουργήσει νέα νομοθεσία όπως και έγινε. η οποία να βελτιώσει την ευελιξία και την ε, πρόσβαση στην απασχόληση των γυναικών. η ανεργία δυστυχώς αυξήθηκε παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για μείωσή της. Υπήρξαν ε, προγράμματα τα οποία εισήχθησαν, φορολογικά μέτρα, φορολογικές ελαφρύνσεις για εκείνους όπου έχουν ακόμα μεν ε, δουλειά όμως βρίσκονται σε πολύ επισφαλή θέση προσπάθησαν να δημιουργηθούν ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας με χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, να δημιουργηθούν επίσης νέες θέσεις εργασίας πιο φιλικές προ ε, τι εργαζόμενες μητέρε και διάφορα άλλα προγράμματα τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Μαριάν Βασίλειεφ από το Ρουμανικό Κοινοβούλιο, από τη Γερουσία μάλιστα. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για το σημερινό συνέδριο. Θα ήθελα να παρουσιάσω την ομιλία μου στα ρουμανικά, στη γλώσσα μου. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω εδώ. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι δεν θέλω να σας ε, φορτώσω με αριθμούς, με στατιστικές και με τεχνικά στοιχεία, αλλά να σας πω δύο λόγια τα οποία έρχονται από τα βάθη της καρδιάς μου, διότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και... να σας πω ότι είμαι μέλος της Γερουσίας από το κόμμα με επικεφαλή στον κύριο Λιακουνέσκου. Και μπορώ να πω ότι στη Ρουμανία υπάρχει μία κοινωνική απογοήτευση. Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο ασχολείται έντονα με το θέμα και τα προβλήματα. Είναι ένα κόμμα το οποίο το οποίο επικεφαλής είναι γυναίκα, το οποίο εκπροσωπείται από πολλές γυναίκες. Και να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια γυναίκες ήταν εκείνες στις ε, σημαντικές και ηγετικές θέσεις του κόμματος. Φυσικά είχαμε και εμείς τα προβλήματά μας, όμως δεν θα σας μιλήσω για αυτό. Το, θα σας μιλήσω για το πρόβλημα των διακρίσεων που αντιμετωπίζουμε στη χώρα. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ίδρυση του κόμματός μας. Και να πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 30% ε, των βουλευτών Έχουμε πάνω από 30% γυναίκες βουλευτές. Για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη χρειάζεται να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες... Ναι, μιλάτε πολύ γρήγορα, λέει η Πρόεδρος. Πράγματι πρέπει να τελειώσω, πρέπει να μιλήσω εντός των ορίων του χρόνου μου. Είναι όμως πολύ δύσκολο, λέει η Πρόεδρος, για τους διερμηνείς αυτό. Σας ευχαριστώ. Όπως έλεγα, τρόποι εξόδου από την κρίση. Ανεξάρτητα από τη μορφή της κρίσης πρέπει να αυξηθεί ο ρόλος των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό χρειάζεται νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ελάχιστη αντιπροσώπευση των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια. Οι γερουσιαστές της Ρουμανίας θα υποβάλουν τις προτάσεις τους για αυτό το θέμα και ελπίζω να έχουμε τη στήριξη και των άλλων ε, πολιτικών κομμάτων πέραν του δικού μου. Στη Ρουμανία θέλουμε να συνεχιστεί η διαδικασία ένταξης, η διαδικασία ολοκλήρωσης και επίσης αυτό περιλαμβάνει και, την, ε, και το Σέγγεν. Ο λαός της Ρουμανίας επιθυμεί την πρόοδο, τη μελλοντική πρόοδο και στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις γυναίκες, τις μητέρες, τις αδελφές. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στην Άννα Πίεσαλ. Ρουμανή και αυτή, από το άλλο νομοθετικό σώμα της Ρουμανίας. Μην διαβάζετε επιγόντως και τηρήστε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η κατάσταση, τα μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση στην Ουρμανία δεν οδήγησε σε οικονομική ανάπτυξη ούτε στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό χρειάζεται η κοινωνία και αυτό χρειαζόταν και αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Η κοινωνική κατηγορία που επηρέαζεται περισσότερο από την κρίση ήταν οι γυναίκες που έχασαν τις θέσεις εργασίας τους, που δεν μπορούν να βρουν δουλειά που τραγικά έχουν σοβαρές δυσκολίες στο να τηρήσουν, να μείνουν στη δουλειά τους. Η οικονομική κρίση αυτή τάραξε σκληρά την ε, ρουμανική οικογένεια και είναι πραγματικά δύσκολο να συνδυάσει κανείς την ε, ε, επαγγελματική με την προσωπική οικογενειακή δουλειά. Η βία για την οποία μιλάμε δεν είναι μόνο η φυσική αλλά και, και, η ψυχολογική βία και οι γυναίκες πρέπει να ζήσουν σε αυτό το βίαιο περιβάλλον όπου πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται ε, καταχρήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν διακρίσεις ε, στην αγορά εργασίας ε, και στην πρόσβαση και στη διατήρηση των, ε, της δουλειά τους. Η νέα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Βίκτορ Πόντα προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα. Εγώ είμαι βουλευτής, μέλος της Κάτω Βουλής και δούλεψα για να διαμορφήσω έναν νέο νόμο που θα υποβληθεί την άλλη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, που έχει με στόχο να αλλάξει την νομοθεσία για την ισότητα ευκαιριών στην Ρουμανία. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κλείσω λέγοντας ότι η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που εκπροσωπώ εδώ ετοίμασε μια γνωμοδότηση για τη στρατηγική για τη διακίνηση ανθρώπων 2012-2016 και για νέα νομοθετικά κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Κύπρου, κ. Φυτής, έχει το λόγο. Ε, με ιδιαίτερη χαρά σας προσφωνώ σε αυτήν τη συνάντηση για ένα τόσο κρίσιμο θέμα που θα μας προβληματίζει όλους. Συγχαίρω την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φίλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία της. Επιτρέψτε μου επίσης να συγχαρώ τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης δεν είναι ουδέτερος από τη σκοπιά του κοινωνικού φύλου. Λόγω των στερεότυπων αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων και των προκαταλήψεων που επικρατούν για το ρόλο και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, οι γυναίκες καθίστανται περισσότερο ευάλωτες από τους άντρες και πλήθονται εντονότερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Εξάλλου, η επιβολή μέτρων λιτότητας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τρόικα έχει οξύνει περαιτέρω το πρόβλημα. Παράλληλα, η αποδυνάμωση πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας οι περικοπέ στα κοινωνικά επιδόματα και στο δημόσιο προπολογισμό στα πλαίσια τη υλοποίηση μέτρων λιτότητα επηρεάζουν το δημόσιο τομέα και κατ' επέκταση τι γυναίκε, οι οποίε κατά πλειοψηφία στελεχώνουν το δημόσιο τομέα. Στα πλαίσια αυτή τη παρέμβασή μα, θα σα ενημερώσω για τι βέρτιστε πρακτικέ και τα μέτρα που υλοποιεί Κύπρος ένεκα τη οικονομική κρίση σε συντομία για τη διευκόλυνση της ένταξης και επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ενδυνάμωση του ρόλου τους. Η ενδυνάμωση λοιπόν των γυναικών συγκαταλέγεται ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυπριακής κυβέρνησης καθώς και οι τομείς της απασχόλησης της οικονομίας καθιστούν τους κύριους άξονες του σχεδίου δράσης για την ισότητα ανδρών και γυναικών 2007-2013 περιλαμβάνοντας σωρία δράσεων με στόχο την ένταξη των γυναικών στην απασχόληση και την οικονομική ενδυνάμωσή του. Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος γνώρισε την ταχύτερη αύξηση ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανόν μαζί με την Ισπανία. Συγκρίνοντας τα ποσοστά ανεργίας στην περίπτωση της Κύπρου, διαπιστώνουμε ότι η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των φύλων μειώθηκε αισθητά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό ανεργία των ανδρών το τρίτο τρίμηνο του 2012 ήταν 12,3% και των γυναικών 11,8%, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών έφτασε το 25,6% στους άνδρες και 27,1% στις γυναίκες. Μέτρα εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, από το Κέντρο Παραγωγικότητας μέσω του Σχεδίου Χορηγιό για Ένταξη στην Απασχόληση με Βέλεκτες ρυθμίσεις και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και τέταρτον, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιεί δύο σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που τονίσατε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τώρα δίνω μέσω το λόγο σε ένα υποψήφιο κράτος μέλος την, και μια εκπρόσωπο, την κυρία Τόπρακ από την Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, λέει πρόεδρος, πλησιάστε το μικρόφωνο σας. Δεν ακούγεστε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να τονίσω ορισμένα περίεργα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης όσον αφορά τη θέση των γυναικών. Τι εννοώ δηλαδή με αυτό. Κατά τη διάρκεια της κρίσης αυξάνεται η ζήτηση γυναικών στην αγορά εργασίας και αυτό διότι πολλές φορές δεν αρκεί ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια και πολλές φορές αυτό οδηγεί και στην ε, αύξηση επίσης των διαζυγίων διότι αυτό δημιουργεί ενδοοικογενειακά προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν από τη μία η αύξηση στην ε, ζήτηση, στην απασχόληση, από την άλλη υπάρχει και η μείωση των ε, ελεύθερων θέσεων εργασίας. Οι γυναίκες στις υψηλόβαθμες θέσεις συνήθως είναι οι πρώτες που θα απολυθούν. Αυτό που τόνισε και η ο Καθέιν εξάλλου. Και μπορεί να σας το πει και η ίδια καλύτερα. Από την άλλη, στα, ε, στις χαμηλόβαθμες θέσεις προτιμούνται από τους εργοδότες οι γυναίκες, διότι οι γυναίκες είναι πρόθυμες να δουλέψουν η μια απασχόληση και τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πολύ λιγότερη εργασιακή ασφάλεια και πολύ λιγότερη κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική ασφάλιση. Δεδομένου, δεδομένου λοιπόν αυτών των ε, συνθήκων στην αγορά εργασίας ή για τις γυναίκες, το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θα έπρεπε να κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κατά ε, το πρόβλημα μέσω του mainstreaming ε, και έχοντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν με μέσω οικονομικής κρίσης μια οικονομική ανάπτυξη. Να σας πω ε, επίσης ότι στο το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ε, στο οποίο ανήκω, στο, ότι μάλλον είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας. Ευχαριστούμε. Μία εκπρόσωπος της πολωνικής γερουσίας, δεν θα τολμήσω να προφέρω το όνομα, η κυρία Μοζανόφσκα. Συγγνώμη γιατί η προφορά μου ήταν φρικτή. Μα δεν πειράζει κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γυναικών του Κοινοβουλίου για την ε, διακοινοβουλευτική αυτή συνάντηση που οργανώσατε και που δείχνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να βρουν μια λύση στην κρίση διότι το... οι δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες ως επιχειρηματίες είναι πολύ μεγάλες. Τονίζω ότι σε ό,τι αφορά το δυναμικό των γυναικών ο στόχος είναι η ισότητα των δικαιωμάτων για να αναδείξουμε τι δυνατότητες έχουν οι γυναίκες. Πρέπει να έχουν την ικανότητα ασφάλειας σε κάθε κομμάτι της ζωής τους, στην ιδιωτική, οικογενειακή ζωή. Ο στόχος είναι να παράσχουμε ασφάλεια και να επιτρέψουμε στις γυναίκες να ε, συνδυάσουν ε, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Σε ό,τι αφορά την συνδιαλλαγή μεταξύ του ρόλου της γυναίκας ως ε, εργαζόμενης και της ιδιωτικής ζωής, είναι κρίσιμο να υπάρξει μια τέτοια ισορροπία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε τους άνδρες που μίλησαν σήμερα, διότι υπογραμμίζουν την ανάγκη εταιρική σχέσης και συνεργασίας χωρίς υπερβολική ε, θηλυκοποίηση σε εισαγωγικά. Η κυβέρνηση της παίρνει μέτρα για την διευκόλυνση της ε, λειτουργίας των γυναικών στην αγορά εργασίας, τους παρέχει καινοτόμα εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι γυναίκες είναι το 46% του ενεργού εργατικού δυναμικού. Υπάρχει πάντα η μισθολογική διαφορά, αλλά σκεφτόμαστε ευέλικτες ε, λύσεις, όπως ε, μη σταθερά ωράρια, τηλεεργασία, το μας απασχολούν τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες, της εταιρικής ευθύνης, της σημασίας των, ε, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και την προστασία των γυναικών των επίτοκων γυναικών και των γυναικών άνω των 50. Ο στόχος είναι η κοινωνική ανάδειξη των γυναικών και σε τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Πρέπει να τηρήσουμε τα ωράρια αγαπητοί συνάδελφοι, γι' αυτό επιμένω. Η κυρία Καζάκα από την Λετωνία έχει το λόγο τώρα. Καλημέρα σε όλους εκπρόσωπο το Κοινοβούλιο της Λετωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα είμαι σύντομη. Καταρχάς ευχαριστώ όλους σας για τις προτάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την παρουσία των γυναικών στον τομέα των επιχειρήσεων. Βέβαια πρέπει να δούμε όμως και πώς πρέπει να ε, ε, ενισχύσουμε την παρουσία των γυναικών στην πολιτική. Θα σας παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία για τη συμμετοχή των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια. Στην Λετωνία έχουμε 23% ε, βουλευτές γυναίκες στο Κοινοβούλιο και 29% γυναίκες υπουργού στην κυβέρνηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίστοιχα έχει 35% γυναίκες και 33% γυναίκες υπουργοί στις εθνικές κυβερνήσεις. Επίσης, να σας φέρω το παράδειγμα ε, της Φιλανδίας, της ε, γειτονικής μας χώρας στο Βορρά. Οι γυναίκες στην ε, Φιλανδία ψηφίζουν εδώ και 100 χρόνια και μόνο τώρα το 50%, υπάρχει 50% συμμετοχή των γυναικών στο κοινοβούλιο ως προϋπόθεση καθώς και στην κυβέρνηση. Χρειάστηκε δηλαδή η Φιλανδία 100 χρόνια χωρίς την εισαγωγή υποχρεωτικής ποσόστοσης για να καταφέρει αυτό το αποτέλεσμα. Πώς θα ε, θεωρούσατε εσείς μια υποχρεωτική ποσόστοση για τα επόμενα δέκα χρόνια ως ένα προσωρινό μέτρο, ως μια μορφή σύστασης προς τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ που ε, θίξατε και αυτό το ζήτημα. Η κυρία Χερκαλκαρά από την Τουρκία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαίρω τις ομιλήτριες. Ε, η ευρωπαϊκή κρίση δεν έπληξε ε, την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια το τουρκικό κοινοβουλίο εισήγαγε μέτρα για να προωθήσει την ε, απασχόληση ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των θέσεων απασχόληση. Η έμφυλη κατάρτιση του προϋπολογισμού που είναι η αρμοδιότητα της Υποεπιτροπής για την Ισότητα των Δύο Φυλών άρχισε να λειτουργεί στι 15 Νοεμβρίου του 2012. Μέχρι στιγμής 13 συνεδριάσεις είχαμε. Η επόμενη έχει προγραμματιστεί για την 20 και 21η Μαρτίου στο Κοντζάιλι. Μεταξύ άλλων θα θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για τις δημόσιες υπηρεσίες τους ΟΤΑ και τις ΜΚΟ που θα εκδοθούν μετά το πέρας των εργασιών της Χάρη στο νέο νόμο της 25ης Φεβρουαρίου 2012 η άδεια μητρότητας αυξήθηκε στις 16 εβδομάδες και η γονική άδεια που ισχύει και για τις γυναίκες και τους άντρες για 24 μήνες άδεια άνευ αποδοχών εισήχθη επίσης στην νομοθεσία. Ε, εν τέλει... Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Κάρμεν Καντανίλα, διότι συνεργαζόμαστε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση και την Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διακριτικής Μεταχείρισης ε, κατά των γυναικών. Ε, συμφωνώ μαζί της, δηλαδή μας μίλησε για τα ψυχολογικά προβλήματα, την κατάθλιψη, φερρυπίν, που θα εκδηλωθούν στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη και να καταπολεμήσουμε ναι μεν τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά προβλήματα αλλά και τα προβλήματα που θα πλήξουν την οικογένεια, την παιδεία, ε, την ανατροφή των παιδιών. Ε, ούτως ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις, όμως ε, με αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα θα έχουμε καταστροφικές επιπτώσεις στο μέλλον. Ιδού. Ε, πρόεδρος, σας ευχαριστούμε για τις μαρτυρίες σας. Ε, ακούσαμε εκπροσώπους χωρών από ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης ε, να χαιρετήσω τους συναδέλφους βουλευτές του Κοινοβουλίου που συμμετέχουν σε εργασίες μας σήμερα και για να ολοκληρώσουμε την πρωινή συνεδρία θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο Γκούσταυσον. Um, θα περάσουμε τώρα στο τρίτο πάνελ. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, στηρίξει τα κράτη-μέλη για να ε, προστατεύσουν τις γυναίκες σε αυτή την περίοδο κρίσης. Θα ακούσουμε τώρα με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και θα στήριξη τις γυναίκες. Ε, έχουμε και στην Επιτροπή Γυναικών ένα σχέδιο έκθεση πρωτοβουλίας για αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας δείξουμε ένα βίντεο. Ο Επίτροπος Άντερ δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, αλλά έκρινε ότι είναι τόσο σημαντικό το ζήτημα που ήθελε τουλάχιστον να περάσει ένα μήνυμα έστω και εξ ε, θα δούμε λοιπόν ένα βίντεο με την παρέμβαση του Επιτρόπου και στη συνέχεια ε, θα ε, συνεχιστεί η συζήτηση. Ελπίζω να είναι όλα ρυθμισμένα όπως πρέπει, τα μάτια στις οθόνες και παρακολουθούμε το βίντεο. It will Υπομονή και έρχεται. Vice Chair, honorable members, ladies and gentlemen, I extend my... Αντιπρόεδρε, Αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι, σα καλωσορίζω θερμά όλου, ιδιαίτερα τι γυναίκε αυτή τη σημαντική ημέρα. Λυπάμαι που δεν μπορώ να παρευρεθώ μαζί, να, εδώ μαζί σα σήμερα, όμω, εκτιμώ την ευκαιρία που μου δώσατε να σα μιλήσω έστω και με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα είναι μία μέρα προβληματισμού για να δούμε πώς, πού έχουμε φτάσει όσον αφορά την ισότητα των φίλων, ιδιαίτερα στον τομέα τη απασχόληση. Και το λέω αυτό διότι η ένταξη στην αγορά εργασία είναι επίση ένα από του καλύτερου τρόπου συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο ένα θεμελιώδε δικαίωμα. Είναι επίση ζωτικό για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα των ε, οικονομιών στην Ευρώπη. Με τη γύρανση του πληθυσμού, με, το, με την πτώση των, ε, του αριθμού των γεννήσεων και με την ε, μείωση, την μελλοντική μείωση των δεξιοτήτων, η εκμετάλλευση όλων των ταλέντων, όλων των ανθρώπων και η ισότητα των φίλων ως παράγοντας ανάπτυξης είναι πιο σημαντική από ποτέ. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον τρόπο που η κρίση έχει επηρεάσει την ισότητα των φύλων. Όταν η κρίση άρχισε το... και οι διαφορές στην απασχόληση ανάμεσα στα δύο φύλλα μειώθηκαν, διότι η κρίση κυρίως επηρέασε τομείς όπως τον κατασκευαστικό και την αυτοκινητοβιομηχανία όπου ε, απασχολούμενταν κυρίως άντρες. Από τότε όμως οι, δαπα... οι περικοπές στις θέσεις εργασίας του δημοσίου και οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες φαίνεται πως είχαν ένα πολύ μεγάλες αρνητικές ε, επιπτώσεις ιδιαίτερα ως προς τις ε, γυναίκες και αυτό οφείλεται ε, ως ένα ε, βαθμό το γεγονός ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στον δημόσιο τομέα και επίσης εξαρτώνται περισσότερο ε, σε ορισμένες υπηρεσίες και στην πρόσβαση τους σε αυτές όπως, για παράδειγμα η παιδική μέρημνα, η μακροχρόνια περίθαλψη και η υγειονομική περίθαλψη. Για να επιτύχουμε τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και την μείωση της φτώχειας πρέπει να, ενισχυθεί, να ενισχυθούν τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των γυναικών. Όμως κοιτάξτε τα νούμερα. Το 2011 το ποσοστό απασχόληση για του άντρε στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών ήταν 70,1% και οι γυναίκε αντίστοιχα 58,5%. Επίση, ένα στου 10 άνδρες εργαζόταν σε ήμια απασχόληση, όμω ο μέσο όρο των γυναικών ήταν πολύ μεγαλύτερο. Τρει στι δέκα γυναίκε εργαζόταν σε ήμια απασχόληση. Η ήμια απασχόληση μπορεί να είναι μια επιλογή, όμω πολλέ φορέ ε, έχει άμεση σχέση με ε, λιγότερες ε, απολαβές ε, ώρα με λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης, λιγο, μικρότερη ε, ασφάλεια και μειωμένη μια μειωμένη σύνταξη. Αυτό κυρίως οφείλεται στις, στις απλήρωτες εργασίες των γυναικών στο σπίτι, στον οικοκυριό, στην παιδική μέρημνα. Επίσης, οι, οι επιπτώσεις στις νέες γυναίκες είναι μεγάλες. Πολλές, η, η, κρίση ενδέχεται ε, να εμποδίσει τις γυναίκες να, να απολαμβάνουν τα πλήρη, ε, τις πλήρης ε, παροχές εμιτρότητας και αυτό μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις ε, των γυναικών όσον αφορά το να κάνουν οικογένεια. Επίσης υπάρχουν και άλλοι ε, πολύ σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εκτός ε, από την ε, κατάσταση στην απασχόληση και αυτοί οι παράγοντες τονίζονται στην έκθεση δύο πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών. Όπως είπε η κυρία Μωρήν Σαρτιέ, η συγγήτρια, οι εργασιακές συνθήκες των γυναικών έχουν γίνει όλο ένα και πιο επισφαλείς και το εισόδημά τους έχει μειωθεί σημαντικά. Αυτό, αυτό οφείλεται στο ε, κενό, στη διαφορά τη μισθολογική ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες και, στο, και ως αποτέλεσμα στην έλλειψη ισότητας στις, ε, στα επιδόματα ανεργίας και στην αύξηση ε, της ε, υποχρεωτικής ημιαπασχόλησης και του αριθμού των, των προσωρινών ή ε, ορισμένου χρόνου εργασιών. Επίση, κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, οι δεξιότητε. Ε, παρότι οι γυναίκε είναι καλύτερε από του άντρε, σε σχεδόν όλου του κλάδου ε, στι χώρε του ΩΣΑ, Πολλέ φορέ οι απόφοιτοι, οι γυναίκες απόφοιτοι στους κλάδους τη επιστήμης, τη τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών είναι πολύ χαμηλός. Και οι γυναίκε που καταφέρουν να αποφοιτήσουν από αυτού του κλάδου, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασία, πολλέ φορέ επιλέγουν να μην εργαστούν στου τομεί αυτού. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα νωρί με τη σχολική εκπαίδευση και τα συστήματα κατάρτιση και να δώσουμε περισσότερε δυνατότητε μαθητεία στι νέε γυναίκε. Κυρίε και κύριοι, τέτοιοι παράγοντε όπω η προσωρινή εργασία, η μεαπασχόληση, οι μονογονεϊκέ ε, οικογένειε, τα μισθολογικά κενά και οι ε, διακοπέ ε, στην εργασία λόγω μητρότητα μπορούν να μα βοηθήσουν να καταλάβουμε γιατί υπάρχουν 12 εκατομμύρια περισσότερε γυναίκε από ότι άντρε που ζουν στη φτώχεια βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η πρόνοια και οι ε, κοινωνικές παροχές είναι οι πρώτοι ε, τομεί ε, στους οποίους γίνονται περικοπές και αυτό οδηγεί σε περισσότερη ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα οι κοινωνικές δαπάνες πρέπει να, πρέπει να θεωρούνται όχι ως κάτι που μπορούμε να περικόψουμε, αλλά ως μια κοινωνική επένδυση. Και αυτό είναι ένα από τα μηνύματα τα οποία προσπαθήσαμε να περάσουμε με, όταν ε, ψηφίσαμε πριν από δύο εβδομάδες το ε, πακέτο κοινωνικών επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πρόοδο των κρατών μελών για την στην ισότητα των φύλων μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εννέα κράτη-μέλη έλαβαν ε, συγκεκριμένε συστάσει αναχώρα όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την επίτευξη καλύτερη ισορροπίας ανάμεσα στην οικογένεια και στην ε, εργασία. Ορισμένες, ορισμένες συστάσεις αφορούν την παροχή επαρκή ε, και οικονομικής ε, φροντίδας ε, παιδικής εμέρινας και ορισμένες άλλες αφορούν την καλύτερη δημοσιονομική αντιμετώπιση των γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει προσδώσει περισσότερη προστιθέμενη αξία στην ισότητα των δύο φίλων στα κράτη-μέλη. Και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο δίνει μεγάλες δυνατότητες ενίσχυσης της ισότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που επετέφθη το Δεκέμβριο στα πλαίσια του ε, ανεπίσημου τριμερούς διαλόγου. Η συμφωνία αυτή προϋποθέτει μία υποχρέωση για καλύτερο ε, mainstreaming και, τα, την υποχρέωση των κρατών μελών να ενσωματώσουν την έμφυλη διάσταση και στις πολιτικές τους και στα προγράμματα που υποστηρίζονται από το Κοινωνικό Ταμείο. Κυρίες και κύριοι, στόχος της ο στόχος της πλήρους ισότητας μπορεί να μας φαίνεται οφθαλμαπάτη, όμως η ανάπτυξη και η ευημερία για το μέλλον θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το πόσο επιτυχείς είμαστε στο να χειριστούμε τα, και να χρησιμοποιήσουμε τα ταλέντα όλων, ιδιαίτερα των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να τον ευχαριστήσουμε προσωπικά γιατί δεν είναι εδώ, αλλά εκτιμούμε πολύ το μήνυμα που μας έδωσε, πολύ σημαντικό για εμάς. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Επίτροπο. θα προχωρήσουμε στην ανάλυση το τι έκανε με την έκθεση ιδίως πρωτοβουλίας επί Επιτροπή Γυναικών. Αυτό που ανέφυγε ο κ. Σάντος στην ομιλία του. Η συγκίτρια έκανε πολύ καλή δουλειά. Φανταστείτε ότι δεν είναι το ευκολότερο πράγμα να μιλάς για οικονομικά θέματα από την αριστερά και την δεξιά γιατί δεν συμφωνούν εν γέννη σε θέματα. Η, η ωστόσο κατόρθωσε να βγάλει ένα ενιαίο πλαίσιο, ένα κοινό πλαίσιο συζητήσεων ε, στην Επιτροπή. Δεν θα πω περισσότερο, θα τη δώσω το λόγο να τα πει η ίδια γιατί έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά σε μια έκθεση που πιστεύω ότι έχει πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω καταρχάς ότι στο έργο αυτό όλες οι πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο και όλοι οι σκιώδεις εισηγητές ε, πρέπει να λάβουν τις ευχαριστίες σας, γιατί δεν θελήσαμε το θέμα αυτό να μας διχάσει. Θελήσαμε το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί ως ένα πολιτικό, κοινό πολιτικό ζήτημα. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που, ανέφε, που είχαν και αυτή τη διάσταση στο μυαλό τους στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι η κρίση, δεν μπορεί, η κρίση των γυναικών και η αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί, δεν πρέπει να αποτελέσει προνόμιο μιας ομάδας. Είναι ένα κοινό πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ό,τι κάνατε, ούτως ώστε στην Επιτροπή Γυναικών, την Επιτροπή μας να έχουμε αυτή τη σφαιρική προσέγγιση και την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια θα έχουμε την ψηφοφορία που θα δείξει αν καταφέραμε τελικά αυτό το στόχο. Το πρώτο που θέλω να τονίσω για τη δουλειά είναι η μέθοδος. Ακολουθήσαμε μία διπλή μέθοδο μέσα στον χρόνο. Πρώτα, την ανάλυση της κατάστασης, την αντιπαραβολή διαφόρων πολιτικών, διαφόρων τύπων πολιτικών για να υπάρξει ένα πρώτο μια πρώτη συνένεση στην Επιτροπή Γυναικών στην αρχή και στην Ολομέλεια κατόπιν, την άλλη τρίτη πιο συγκεκριμένα. Η δουλειά μας που θα είναι και προσβάσιμη online επικυρώθηκε από μια στατιστική μελέτη που της οποίας χθες ε, δώσαμε τα πρώτα αποτελέσματα Εν τέλει μεταξύ της μεθόδου ανάλυσης και της στατιστικής, συνδυάζοντας την μεθοδική ανάλυση και την ε, ε, στατιστική ανάλυση είχαμε κοινά, ε, κοινή δουλειά, είχαμε κοινά αποτελέσματα. Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι η κρίση, ο αντίκτυπος της κρίσης απλά μεγεθύνει προϊφιστάμενα προβλήματα. Ξέρετε, συχνά σε πολλές χώρες η, η καλή οικονομία έκρυβε τα προβλήματα και κανείς δεν πια τα χτυπήσει. Παράδειγμα, οι μισθολογικές αποκλήσεις μεταξύ ανδρών γυναικών. Η μερική απασχόληση, όπου οι γυναίκες ήταν κυριαρχούσαν. Τα προβλήματα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, όπου οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες. Έχουμε στατιστικά χώρα προς χώρα, μπορεί να τα δείτε και θα διαπιστώσετε και συνολικά στην Ευρώπη και σε κάθε χώρα τα αποτελέσματα. Όλα αυτά τα θέματα, μερική απασχόληση, το τόσο χαρακτήρα των θέσεων εργασία, υπήρχαν και οι γυναίκε ήταν κυρίαρχε παντού σε όλα αυτά τα προβλήματα. Η κρίση ήρθε να χτυπήσει αυτή την, αυτό τον έφραυστο χαρακτήρα των γυναικών στη δουλειά, στη θέση των χώρο εργασία, που τον επιδίνωσε γιατί αύξησε την οικονομική αύξησε, αυξήθηκε, αυξήθηκαν τα ζητήματα λόγω της υπολογικής κρίσης. Τι έχει κρίση, μερική απασχόληση, συμβάσει συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αβέβαιες θέσεις εργασίας, όλα αυτά η οικονομική κρίση τα ανέδειξε. Τρίτον, συζητήσαμε πολύ πολιτικά στο Συμβούλιο ιδίως και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέγοντας εγώ θέλω λιτότητα, έλεγε ο εγώ θέλω ανάπτυξη, έλεγε ο άλλος. Αυτές οι συζητήσεις είναι ξεπερασμένες. Πρέπει ταυτόχρονα να μπορούμε να κάνουμε σωστές πολιτικές μείωσης της υπερχρέωσης των κρατών και πολιτικές ανάπτυξης ταυτόχρονα. <clears throat> Γιατί όπως είπε προηγουμένως ο Επίτροπος κ. Άντορ, η οικονομική και κοινωνική υγεία της Ευρώπης περνάει από τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασία. Και δεν θα έπρεπε να δημιουργούμε διπλές στρατηγικές. Θα έπρεπε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε, όπως μαζί το κάναμε πρόεδρε στο ζήτημα αυτό, μία πολιτική που θα επιτρέπει ταυτόχρονα αυτή τη διπλή προσέγγιση. Τα σημεία που μένουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί είναι τρεις μηχανισμοί που δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθούν. Πρώτο εργαλείο. Μείωση των μισθολογικών αποκλήσεων ανδρών γυναικών. Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η μισθολογική διαφορά τη στιγμή της πρόσληψης μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας είναι περί το 17%. Και θα πρέπει να προσθέσω ότι η γυναίκα με την κρίση μπαίνει πιο αργά στην αγορά εργασία, παρότι έχει περισσότερες θέσεις εργασίας, από, περισσότερα πτυχία από ότι ο, άνθρωπος, ο άνδρας. Αυτή η μισθολογική απόκληση που είναι απαράδεκτη αυξάνεται περαιτέρω κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής της γυναίκας. Κάθε γέννηση παιδιού, μετά από, αυτό είναι μελέτη του ΩΣΑ, σε όλες τις χώρες δείχνει ότι κάθε γέννηση παιδιού μειώνει κατά 12%, αντιστοιχεί με μείωση 12% του μισθού του άντρα σε σχέση με το μισθό της γυναίκας. Γιατί? Διότι από τη γέννηση του πρώτου παιδιού και μετά η γυναίκα έχει την τάση να ζητάει θέσεις με μικρότερη ευθύνη για να ασχοληθεί με το μωρό. Ενώ ο άντρα θα πάρει μία θέση με μεγαλύτερες ευθύνες. Αμέσως, αμέσως μεγαλώνει το χάσμα. Κάθε γέννηση παιδιού θα συνεχίσει αυτή την επιδείνωση. Καλή, καλή 12% κάτω. Στο δεύτερο παιδί η γυναίκα πολύ συχνά θα μπει σε ένα μερική απασχόληση 80%. Πολύ συχνά οι γυναίκες που έχουν τρία παιδιά κατά μέσο όρο δουλεύουν 50% του χρόνου τους. Βλέπετε λοιπόν ότι το χάσμα μεγαλώνει που σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν πιο ισοπεδωμένες σταδιοδρομίες από τον άντρα. Και αυτό θα το ξαναπώ πρόεδρε όταν ε, δούμε τον κύριο Μπαρόζο και τη Βιβιάν Ρέντιν την άλλη τρίτη. Διότι πρέπει όλοι να χτυπήσουμε την ισοπεδωμένη σταδιοδρομία της γυναίκας. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο αντιμετώπιση των ε, ανισοτήτων αλλά και απελευθέρωση της γυναίκας στην επαγγελματική ζωή. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει πολύ. Διότι όλα τα κράτη-μέλη επενδύουν τεράστια ε, ποσά στην ισότιμη ε, κατάρτιση αγοριών κοριτσιών και οικογένειες. Και σας κοιτώ κυρία μου διότι η δική σας παρουσίαση σε αυτό το θέμα ήταν πολύ σημαντική. Πώς μπορούμε να φανταστούμε να επενδύσουμε για να επιτρέψουμε την ανάπτυξη, την, την, να καρποφορήσει αυτή η επένδυση εάν τη γυναίκα την αφήνουμε μόνο στην, ε, στο να δουλεύει 50% του χρόνου της σε μια ε, διαδικασία που δεν, ε, σε μια σαδιοδομία που δεν εξε, εξελίσσεται. Πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε την κατάρτιση, την ισότητα εργασίας, τη συναδιαλλαγή επαγγελματικής και οικογενειακής καριέρας, τόσο ώστε η γέννηση κάθε παιδιού να μην επηρεάζει αρνητικά την εμπλοκή της γυναίκας στην επαγγελματική της καριέρα και όλοι μαζί να χρησιμοποιήσουμε το μοχλό στα Ξέρετε, όλο αυτή η διαδικασία είναι πολύ σύνθετη και η ευρωπαϊκή πολιτική μέσω και του ευρωπαϊκού εξαμήνου, όπως είπε ο κύριος Άντορ, αλλά και κάθε εθνικό επίπεδο, κάθε κράτος μέλος, με κοινά κριτήρια θα πρέπει να μπορεί να μετρά σε μόνιμη βάση τις συνέπειες των δημοσίων πολιτικών για να μην ξυπνάμε απλά το 2013 και να πούμε τι κάνουμε για τις δημόσιες πολιτικές μετά την κρίση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το πρόβλημα να αναπτυχθεί χωρίς αυτή την δυνατότητα αντίδραση. Σας εφιστώ την προσοχή σε ένα σημείο που μας σώκαρε ιδιαίτερα. Σήμερα, μεταξύ των κριτηρίων πρόσληψης που δείχνει και το Ευρωβαρόμετρο και δεν σας αρέσει περισσότερο τα τρία πρώτα κριτήρια πρόσληψης ε, των γυναικών είναι έχει παιδιά ή δεν έχει. Ένα προσωπικό κριτήριο που διακρίνει με αρνητικό τρόπο, δεν διακρίνει θετικά, ε, αποκλείει. Δεύτερο κριτήριο, διαθεσιμότητα ωραρίου. Γι' αυτό με, με εντυπωσίασε όταν μιλούσατε για τη χρήση της τηλεεργασίας ε, που θα κάλυπτε αυτή τη ε, διάκριση. Και τρίτο, σας το λέω έτσι ομά, αν έχουν ωραίο παρουσιαστικό. Η επαγγελματική εμπειρία είναι το έβδομο κριτήριο πρόσληψης μιας γυναίκας τι γίνεται με τους άντρες. Σε επίπεδο 27 κρατών μελών. Αλλά πηγαίνετε να δείτε τι λέει το καθένα. Πρώτο κριτήριο πρόσληψης, επαγγελματική εμπειρία. Για τη γυναίκα είναι το έβδομο, για τον άντρα το πρώτο. Δεύτερο κριτήριο, προσόντα. Θετικά προσόντα. Τρίτο κριτήριο, διαθεσιμότητα. αυτό που χρησιμοποιούμε αρνητικά για τη γυναίκα το χρησιμοποιούμε θετικά για τον άντρα. Το γεγονός ότι ένας άντρας έχει ή δεν έχει παιδιά είναι το δέκατο στη σειρά κριτήριο για τον άντρα ενώ είναι το πρώτο, το δεύτερο για τη γυναίκα, το πρώτο για τη γυναίκα. Η ανάλυση του Ευρωβαρομέτρου δείχνει τι είμαστε δείχνει την κοινωνία στην οποία ζούμε. Και νομίζω ότι όταν διαβάζουμε τα κριτήρια αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα. Άκουσα το πρωί να μιλάμε για την ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων. Και εδώ ωστόσο η κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολη. Να τονίσω κάτι άλλο. Την πυραμίδα των, της δουλειάς. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολυ... μπορούμε να αναλύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές εν ώψη του 14-20. Στην πυραμίδα αυτή και εν ώψη του 2020 ξέρουμε ότι το 15% των θέσεων εργασίας χαμηλού επίπεδου στη βάση της πυραμίδας θα χαθούν. Ότι οι θέσεις υψηλού επίπεδου προσόντων, η κορυφή της πυραμίδας θα αυξηθούν κατά 15%. Δείτε τις διάφορες μελέτες που έχει κάνει το ΣΕΝΤΕΦΟΠΡΟ το ΣΕΝΤΕΦΟΠ στη Θεσσαλονίκη. με το οποίο συνεργαζόμαστε στενά. Είδατε, το είπαν πολύ σήμερα το πρωί, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στα χαμηλά, στις χαμηλές θέσεις, ενώ είναι λιγότερες στα ψηλά επίπεδα. Αν δεν φροντίσουμε λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση, θα έχουμε το, ως επίπτωση της κρίσης και την ανοικοδόμηση των θέσεων εργασίας μετά την κρίση που θα απαιτήσει μία νέα διαμόρφωση προσόντων των μισθωτών εν γέννη, μέσα στην οποία αναδιαμόρφωση δεν θα προχωρήσουν με ταχύτερο ρυθμό οι γυναίκες. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να έχει διορθωτικές πολιτικές και επανέρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Άντερ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει φτιαχτεί για να προλαμβάνει τέτοια προβλήματα. Σας παρακαλώ κινηθείτε σε κάθε κράτος ώστε η επιστροφή των γυναικών στο χώρο εργασίας, η επικύρωση των ε, εμπειριών, των, ικανοτήτων, των ικανοτήτων, η μόνιμη ε, κατάρτιση να είναι εποφελής ευρέως για τις γυναίκες, κάτι που θα διορθώνει την υφιστάμενη τωρινή κατάσταση. Προφανώς κάτι ξέχασα να σας πω. Η μισθή για τις γυναίκες είναι χαμηλή. Η απασχόληση είναι λιγότερο ασφαλής. Άρα η κρίση έχει μία επίπτωση που είναι μια ήσυχη επανάσταση, μια σιωπή επανάσταση. Φεύγει η γυναίκα από τη δουλειά μόνη τη. Δεν έχει μεγάλο μισθό, ε, έχει υψηλά, υψηλά, υψηλές υποχρεώσεις παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, άρα φεύγει από την αγορά. Ο αντίκτυπος της κρίσης στην αγορά, αν δείτε τα στατιστικά, δεν είναι τόσο διαφορετικές, διαφορετικός ε, σε άντρες και γυναίκες. Αλλά τι συμβαίνει. Είναι λιγότερο πολυάριθμες. Φεύγουν. Δεν φεύγουν τελείως από τον χώρο αγοράς εργασίας, φεύγουν από τον χώρο αγοράς μισθωτής, αμοιβόμενη εργασίας και δουλεύουν σε δουλειές φιλανθρωπικού χαρακτήρα στις μη, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μη αμοιβόμενε δουλειές. Καταλήγουμε λοιπόν στο να υλοποιούμε πολιτική να υλοποιούμε πολιτικές επιστροφή των γενικών στον χώρο εργασία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για παράδειγμα δουλεύει για το σκοπό αυτό, αλλά μην ξεχνάτε ότι το, Κοινωνικό Ταμείο είναι φτιαγμένο και για τα νέα προσόντα των γυναικών στην αγορά. Άρα το 2014 μόνο αυτές που ήταν στην αγορά εργασία θα μπορούσαν να υποφεληθούν από τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταμείου. Και μιλώ πολύ για το Κοινωνικό Ταμείο γιατί είμαι μόνιμη εισηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα εργαλείο εξαιρετικό για να σας βοηθά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διαμορφώσουμε αυτή την ισότητα ανδρών και γυναικών. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Σας δίνω το λόγο, αλλά βλέπετε ότι έχουμε πολλές μάχες ακόμα να κάνουμε, ανεξάρτητα από τις πολιτικές επιλογές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μάσατη υπάρχουν ε, πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να πει και ακούσαμε ήδη πάρα πολλές παρατηρήσεις. Ε, ξέρω τα γνωρίζουμε όλα αυτά, αλλά ε, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό όταν ακούμε ότι δεν υπάρχει επαγγελματισμός στις προσλήψεις, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη το ότι ο υποψήφιος είναι η γυναίκα, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και ε, επίσης είναι ανησυχητικό το ότι θεωρείται ότι την ε, μεγαλύτερη ευθύνη για την ανατροφή των ε, παιδιών την έχει η γυναίκα, ενώ χρειάζονται δύο για να γίνει ένα παιδί. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείται πρωτίστως υπεύθυνη η γυναίκα. Αλλά τι ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, ε, κοιτάζω τον κατάλογο μιλητών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, ε, γιατί στις 12.30 η καταπληκτική διερμηνής, λέει ο Πρόεδρος, τον ευχαριστούν πολύ για την ευρωχροσύνη, θα πρέπει να αποχωρήσουν. διότι εργάζονται μόνο για 3,5 ώρες κατά νότα το όριο, λοιπόν, οπότε παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Η κυρία Γκρουμάη θα πάρει πρώτη το λόγο. Ε, είστε και σκιώδης ε, εισηγήτρια για την ε, έκθεση της κυρίας Μοχάν Παρακαλώ, είστε βουλευτής, σας δίνω το λόγο. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως πραγματικά η Ελίζαπεθ μας έδειξε Πώ πρέπει να συμπεριφερόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσει που έχουν πλήξει τις γυναίκες και άντρε. Τώρα θα αλλάξω, θα μιλήσω ουγγρικά γιατί έχουμε εξαιρετικού διερμηνείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελίζαμπεθ έδειξε με την έκθεση αυτή ότι το θέμα αυτό είναι διακομματικό και πρέπει να συζητηθεί διακομματικά από όλες τις κοινοβουλευτικέ ομάδες έτσι ώστε να επιτευχθεί συνένεση, πραγματική συνένεση. Διότι αυτό το συμφέρον, το συμφέρον των γυναικών, το καλό των γυναικών πρέπει να μην έχει πολιτική απόχρωση. Για πάρα πολλούς από εμάς και από εσάς ε, το θέμα της ισότητας των γυναικών είναι κάτι πάρα πολύ ε, κοντινό, είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Η Επίτροπος Ρέντινγκ δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει. Το θέμα αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία διότι η κρίση έχει επιδεινώσει τη θέση των γυναικών. Τα μέτρα λιτότητας έχουν εντείνει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες και έχουν μεγαλώσει και το χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν πληγεί διπλά από την κρίση, από την κρίση και ε, οικονομικά αλλά και ηθικά, διότι αυτή η κρίση είναι και ηθική, ας μην το ξεχνάμε, είναι κρίση αξιών. και έχει επιδεινωθεί και εμέσως μέσω των ε, περικοπών στις κοινωνικές παροχές. Η κρίση αυτή όμως έθεσε επίσης και το ερώτημα της ίσης μεταχείρισης ε, ανδρών και γυναικών. Και με αφορμή αυτό πρέπει να συζητήσουμε το θέμα και να το συζητούμε ολοένα και συχνότερα, να είναι ολοένα και συχνότερα στην ημερήσια διάταξη. Οι ανισότητες, όπως είπα, έχουν επιδεινωθεί και η κρίση πολλές φορές χρησιμοποιείται ως ε, παραπέτασμα καπνού από πολλούς πολιτικούς έτσι ώστε να γίνουν περικοπές στον κοινωνικό τομέα και στις ε, κοινωνικές παροχές. Εμείς ως Επιτροπή Γυναικών έχουμε ως έργο να συζητήσουμε αυτό το θέμα, να το θέτουμε ε, στην ημερήσια διάταξη και να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση αυτή. Μια κατάσταση στην οποία οι γυναίκες είναι υποαπασχολούμενες, έχουν χαμελότερες απολαβές από τους άνδρες και πώς θα βελτιώσουμε την θέση τους. Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο θα ασκεί κριτική και θα είναι σαφές και το μήνυμα αυτό θα περιέχει το ότι πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με την δημιουργία υποχρεωτικών μέτρων. Μέτρων τα οποία θα βάλουν στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει, ε, έχει ζητηθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή και να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Εμείς πρέπει πραγματικά να δώσουμε το πρέπον βάρος στο θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό τι συμπεριλαμβάνει. Συμπεριλαμβάνει μια αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, να σας πω, είμαι η συγγήτρια για μια έκθεση για την πρόσβαση σε κοινωνικές ε, υπηρεσίες και την ε, σωστή εφαρμογή της ε, οδηγίας της αντίστοιχης. Εδώ πολλά κράτη-μέλη έχουν αναλάβει να εναρμονίσουν και να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως δυστυχώς η ευρωπαϊκή κρίση έχει επιβραδύνει την διαδικασία αυτή και η κατάσταση φυσικά ως αποτέλεσμα έχει επιδεινωθεί. Έχει μεγαλώσει τόσο πολύ η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ώστε σε σχέση με τους άντρες οι γυναίκες είναι σαν να δουλεύουν 95 μέρες το χρόνο δωρεάν. πρέπει, και το επαναλαμβάνω αυτό, να θεσπίσουμε υποχρεωτικά μέτρα. Και πρέπει επίσης να εργαστούμε πολύ περισσότερο εντατικά για την ισότητα των ε, ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον, στους ε, τομείς της πολιτικής και ιδιαίτερα στους τομείς της πολιτικής που ασχολούνται με την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Πρέπει πραγματικά να πάρουμε το, τη δουλειά μας στα σοβαρά και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αντιπαράθεσή μας με το Συμβούλιο. Όσο διαρκεί αυτή η κρίση, εμείς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, πρέπει να εξετάσουμε όλα τα στατιστικά στοιχεία, να λάβουμε υπόψη τις επιστημονικές μελέτες και όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άνδρες και οι γυναίκες, περιμένουν εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει ξεκάθαρα βήματα. Ευχαριστώ πολύ, μας τελειώνει ο χρόνος. Τώρα θα περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, την κυρία Καζάκα από την Λετωνία. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και για την ε, συζήτηση και το πάνελ που είχαμε. Η Λετωνία εισήλθε στην κρίση το 2008 και για μας κράτησε τέσσερα χρόνια. Έγινε νέα νομοθεσία για την δημοσιονομική πολιτική. Εφαρμόσαμε και, την, ε, και τις ε, συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταφέραμε να ξεπεράσουμε την κρίση και σύντομα να ταχθούμε και στην Ευρωζώνη. Οι αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε περίοδο κρίση, είναι, κρίσης, είναι κάτι που γίνεται σε περίοδο κρίσης. Όμως, να σας πω ότι το 35% των φτωχών στη Λετωνία είναι παιδιά. Και τώρα εμείς στην Λετωνία ε, δημιουργούμε διάφορες πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε αυτό ακριβώς το πρόβλημα της φτώχειας των παιδιών. Επίσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την διακίνηση ανθρώπων, την ενδοοικογενειακή βία, την μετανάστευση για οικονομικούς λόγους και τα γρήγορα δάνεια, τα οποία πολλές φορές έχουν οδηγήσει πολλές οικογένειες σε χρεοκοπία. Αυτό που θέλω να πω όπως και να έχει, είναι ότι η αντιμετώπιση της κρίσης για εμάς τη Λετωνία, μια χώρα που πρόσφατα επανάκτησε την ε, δημοκρατία, αντιμετωπίστηκε και με ε, πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια. Εμείς ως πολιτικοί, παρότι ε, καλωσορίζουμε την προσέγγιση σας ε, επίλυσης της κρίσης και παρότι καλωσορίζουμε τις ε, πρωτοβουλίες σας για τα δικαιώματα των γυναικών, να πω ωστόσο ότι πάρα πολλές από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις μας αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί σε χρεοκοπία λόγω της ελλειπούς χρηματοδότησης. Επίσης υπάρχει πρόβλημα στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω, να ρωτήσω την Επιτροπή για το πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, τι συστάσεις μπορεί, μπορούν να γίνουν για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και το πώς αυτές, η στήριξη σε αυτές μπορεί να βελτιώσει την, την κατάσταση. Επίσης, πρέπει να κατανοήσουμε τα αναπαραγωγικά μας δικαιώματα, τα οποία αμφισβητούνται τον τελευταίο καιρό και παρατηρείται μία τάση οπισθοχώρησης και πισωγυρίσματος για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Ας το λάβουμε αυτό υπόψη. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ ως ε, αποτέλεσμα της ε, κρίσης και να πω ότι στην Λετωνία Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καλύτερες πολιτικές όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια. Αλλά σας παρακαλώ βοηθήστε μας, βοηθήστε μας να γίνουμε μέλος του ΟΣΑ. Αυτό είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας και πιστεύουμε ότι μέσω της χρήσης βέλτιστων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να βελτιώσουμε το ζήτημα της ισότητας στην χώρα μας. Να κλείσω λέγοντα ότι Χαίρομαι πάρα πολύ που η Λετωνία είναι 8 χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά ήδη, όμω υπάρχουν εξίσου πολλά στην Λετωνία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία χρήζουν βελτίωση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στον κύριο Πέλες, στην κυρία Πέλε. συγγνώμη. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ουγγρικά. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα είμαι σύντομη, αλλά θα κάνω ότι μπορώ να περιοριστώ στα απολύτως απαραίτητα. Ε, να σας πω ότι δεν είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής, είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και από οικονομική σκοπιά θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω την κατάσταση. Καταρχάς συμφωνώ με αυτά που λέει η συγγήτρια, η κυρία Σαχτιέ. Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση και τη βρίσκω πολύ θετική την προσέγγιση που παρουσιάζεται. Τα γυναίκες είναι θύματα αυτής της κρίσης και έτσι πρέπει να το δούμε, έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ε, όχι μόνο από ευρωπαϊκή σκοπιά, αλλά και από πλευρά κρατών μελών. Μέτρα από τα οποία θα εφαρμόσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν την κατάσταση ε, των γυναικών. Διότι η βελτίωση αυτή είναι προτεραιότητα. Ακόμα και σε περίοδο κρίσης στην οποία, κατά την οποία γίνονται περικοπές. Θα σας ε, αναφέρω ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει επιτύχει ορισμένα αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Όπως σας είπα και η συναδελφός μου προηγουμένως, υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες δεν είχαμε ακόμα αρκετό χρόνο για να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Ο ένας ε, τομέας αφορά τις, ε, την ασφάλιση. Δυστυχώ δεν έχουμε λάβει απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ερωτήματά μα και έτσι αναγκαστήκαμε να του υποβάλουμε για δεύτερη φορά εκ νέου ερώτηση Πώς δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία και η στρατηγική Ευρώπη 2020 έτσι ώστε να συνδεθούν και να προωθήσουν τις ε, γυναίκες επιχειρηματίες. Έπειτα, ένα δεύτερο ερώτημα που έχει προκύψει από αυτά που άκουσα από την εισηγήτρια για το μισθολογικό κενό ε, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Το άρθρο 157 της Συνθήκης της Λισαβόνας αναφέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία μισθολογική διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες και τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να το τηρήσουν αυτό. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τους ελέγχει και γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε μια γραπτή δήλωση Και επειδή είμαι προσωπικά υπεύθυνη για αυτή, θα ήθελα να ζητήσω την στήριξή σας. Με την γραπτή δήλωση αυτή ζητούμε καλύτερο έλεγχο εφαρμογής των ε, κανόνων και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. κλείνοντα να σας ευχηθώ καλή τύχη και καλή επιτυχία στην συνέχιση της δουλειά σα και εύχομαι να καρποφορήσει αυτό πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Οι διεμηνείς μας ενημερώνουν ότι θα φύγουν. σύντομα. Έχουμε δύο ακόμα ομιλητέ. Πρώτα, ο κύριος Μαρσέτη από την Επιτροπή. Θα θέλατε να λάβετε το λόγο. <laughs> That Ρητορικό το ερώτημα. Με συγχωρείτε. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Κουιντανίγια. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή συζήτηση ε, για τη γυναίκα στην οικονομική κρίση. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Η κυρία Σαχτιέ έθεσε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Η τόσο σημαντική αυτή συζήτηση για την οικονομική κρίση που ολοκληρώσετε στην Επιτροπή του Κοινοβουλίου με μεγάλη συνένεση των πολιτικών ομάδων και η συμφωνία να βγει η κρίση, να δείξουμε την, το γυναικείο πρόσωπο της οικονομικής κρίσης είναι θετικό. Θα ήθελα ωστόσο να πω και κάτι άλλο σημαντικό. Είπατε πράγματα που συζητήθηκαν, είπαν πράγματα σήμερα το πρωί, την μισολογική ανισότητα, τον ευάλωτο χαρακτήρα της δουλειάς, τον εξαιρετικά πατριαρχικό τρόπο α, πρόσληψης γυναικών. Είπαν, ε, είπε η ομιλήτρια ή η συγγήτρια ότι ο, η, φυσιογνωμία, ο σωματότυπος είναι το βασικό, ο τρίτος βασικός λόγος πρόσληψης μιας γυναίκας. Εγώ θέλω να πω ότι πολλά χρόνια χρειάζονται για να αναδείξουμε την γυναίκα, για να αναδείξουμε την ισότητα. Σήμερα πρέπει να επανέλθουμε στο να σκεφτούμε ότι η οικονομική κρίση είναι καταστρεπτική για τη δουλειά των γυναικών, ότι η οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει στο ότι εκατομμύρια, χιλιάδες εκατομμύρια γυναικών χάνουν τα δικαιώματα τους. Και ρωτώ κύριε Σαρτιέ, είναι τόσο σημαντική η, η ηγετική θέση του Κοινοβουλίου, όπως και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη στιγμή που διαμορφώνουμε πολιτικές που καθιστούν δυνατό να μην έχει γυναικείο πρόσωπο η οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Κύριε Σαρτιέ τελευταία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για, όλες αυτές τις, ε, για όλα αυτά τα σχόλιά σας. Εγώ θα είμαι γρήγορη και θα προσπαθήσω να κάνω σύνθεση του τι υπόθηκε. Πρώτον, για τα δύο ερωτήματα που τέθηκαν από τους συναδέλφους της Οικονομικής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να συναντήσουμε την, ε, το σκεπτικό και της Οικονομικής Επιτροπής στη δική μας θέση. Ναι, προφανώς πρέπει να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα στις γυναίκες. Και προφανώς αυτό είναι η δουλειά της γυναίκας, είναι ένα βασικό εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσει η γυναίκα να έχει συμπληρωματική κατάτηση που θα της επιτρέπει να πετύχει, διότι και εκεί ε, δεν μπορεί να πούμε ε, γυναίκες πάρτε το, τον τομέα της απασχόλησης χωρίς τίποτα άλλο. Τα δίκτυα είναι σημαντικά ανδρών ή γυναικών, αλλά πρέπει να συνοδεύονται γιατί Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα χωρίς να τις βοηθήσουμε να πετύχουμε. Και η πολιτική της Ευρώπης του 2020 ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί. Δεύτερο θέμα, έχετε δίκιο. Το άρθρο 157 της συνθήκης της Λισαβόνας θέλει να χτυπήσει τις μισθολογικές ανισότητες αλλά ξέρετε ότι πολλά πράγματα περιλαμβάνονται και στην εθνική νομοθεσία για θέματα ισότητας που δεν γίνονται σεβαστά. Και αυτό είναι το χειρότερο. Διότι έρχονται οι συνάδελφοι βουλευτές που λένε το λέει ο νόμος άρα υπάρχει, αλλά αυτό που εμείς ε, θέλουμε είναι όχι μόνο να τα λέει ο νόμος, αλλά και να τα κάνουμε. έχετε δίκιο. Η πρόοδος των γυναικών δεν είναι γραμμική. Είμαι ιστορικός των δικαιωμάτων της γυναίκας και σε κάποιες στιγμές της ιστορίας υπάρχουν μεγάλες καμπές προς τα άνω ή προς τα κάτω. Μην νομίζετε ότι μπορούμε να στήσουμε κάτι στέρεο ή οριστικό. Κάποια στιγμή μπορούμε να πάμε μπροστά, κάποια στιγμή μπορούμε να πάμε πίσω. Η, η χρήση είναι στιγμή ε, αν, επανεξέταση της κατάστασης των γυναικών. Όταν τα κράτη ε, μπαίνουν σε περικοπές των πολιτικών τους, ταυτόχρονα πρέπει να μας οδηγήσουν σε κινητοποίηση, ούτως ώστε η Ευρώπη να λειτουργήσει και ως ε, σταθεροποιητικός παράγοντας. Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι σήμερα συμβάλαμε σημαντικά στις συζητήσεις. Ε, ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν. Το ότι ξεπεράσαμε τον χρόνο είναι καλό πράγμα. Βέβαια δεν είναι δική μου δουλειά, δεν, δεν είναι κάτι το οποίο χαίρομαι να διακόπτω τους φοιτητέ, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία γιατί επέτρεψε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι η συζήτηση μια πολύ καλή συζήτηση με πολύ προοπτική, νέες ε, πληροφορίες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξασφαλίζει ότι η διάσταση του φύλου είναι παρούσα σε όλες τις πολιτικές. Ευχαριστώ και καλό σας μεσημέρι.